Ok, je vous propose de commencer... Ωραία, σας προτείνω να ξεκινήσουμε. Έχετε την ημερήσια διάταξη, υποθέτω ότι μπορούμε να την εγκρίνουμε. Σήμερα έχουμε διερμηνία προς όλες τις γλώσσες, εκτός από τα γοηδελικά και τα κροατικά. Λάβατε τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, της προηγούμενης και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας. Και να ξεκινήσουμε απευθείας την ακρόασή μας. Υπενθυμίζω ότι στις 23 Μαρτίου η Επιτροπή μας έκανε μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό που είναι σημαντικό, κοινωνική προστασία και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με παρουσία της Επιτρόπου Μαριάν Τάισεν που παρουσίασε το σχέδιο αναθεώρησης. Είμαστε σε δημόσια ακρόαση για να εξετάσουμε περαιτέρω τη συζήτηση. Το θέμα αυτό, να το συζητήσουμε περαιτέρω. Και θεωρώ ότι θα βοηθήσει τον ε, εισηγητή μας κύριο Μπάλας και τους Σκιώδης για να συνεχίσουν την εργασία τους επ' αυτού. Θα ακούσουμε τρεις παρουσιάσεις. Από τη μία θα έχουμε την παρέμβαση του δόκτωρα Άιχενχόφα, που είναι πρώην καθηγητής ε, αστικού δικαίου και εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Όσναμπρουκ και το Πανεπιστήμιο της Γένα στη Γερμανία. Κατόπιν θα ακούσουμε την κυρία Ευλίν Ντεγιόγγ που είναι ειδική για θέματα φρολογίας στο γραφείο Ernst Young στο Eindhoven στην Ολλανδία και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Κάρλος Γκαρθία Ντεκορτάθαρ Νευρέδα που είναι αναπληρωτής διευθυντής για τις κοινωνικέ υποθέσεις, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την υγεία και την προστασία των καταναλωτών στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας. Θα δώσω ε, με τη σειρά το, σε καθένα τον λόγο 10 λεπτά και κατόπιν θα ακούσουμε και τον εισηγητή, των σκιωδών και τις ενδεχόμενε ερωτήσεις ή σχόλια. Να δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Άχενχόφερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λειτουργεί το μικρόφωνο. Η πρόταση για την οποία θέλω να μιλήσω στην ουσία ασχολείται με τρία κυρίως θέματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. Καταρχάς, τα τελευταία χρόνια, τέθηκε το θέμα και μέσω της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μάλιστα με οξυμένο τρόπο, τι σχέση έχουν οι διατάξεις για τον συντονισμό των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης. Υπήρξε μια σειρά από πολύ εντυπωσιακέ αποφάσεις που έκαναν εντύπωση δηλαδή οι οποίες ε, έχουν ληφθεί υπόψη για αυτή την πρόταση και αξιοποιούνται για να μεταξελιχθεί το υπάρχον δίκαιο συντονισμού. Υπάρχει μια πρόταση που έχει να κάνει και με το συντονισμό των υπηρεσιών φροντίδας και με μια νέα κατάσταση για την ασφάλιση ανεργίας. Υπάρχουν ε, πολλά άλλα θέματα, αλλά δεν θα ασχοληθώ με αυτά. Καταρχάς για το βασικό θέμα. Κοινωνική πρόνοια και συντονισμός των εργατικών δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μια σειρά από αποφάσεις θεωρεί ότι για τα δικαιώματα κοινωνικής προνοίας για τους μη οικονομικά ενεργούς ε, πρέπει να προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις από τον συντονισμό, ιδιαίτερα για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των πολιτών και από την απέτηση που υπάρχει για να θεωρείται ο τόπος διαμονής ως βασική προϋπόθεση. Αυτό πρέπει ακριβώς να ε, ε ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης που καθορίζει και το άρθρο 24.2. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη πρέπει να προβλέπουν κάποιες εξαιρέσεις στα πλαίσια της ε, ασφάλισης ανεργίας και περίθαλψης. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προσπάθεια της μεταρρύθμισης της νομοθεσίας συντονισμού και υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογική σκέψη που λέει ταξής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μεταδίδει αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη πρέπει να θεωρεί ότι δεσμεύεται ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για τα ανθρώπινα δικαιώματα που, που προκύπτουν από τη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι συμπεριλαμβάνονται και τα κοινωνικά δικαιώματα που θεωρούνται ιδιοκτησία στα πλαίσια του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οπότε δεν μπορούν να παραβιάζονται. Και το θέμα είναι εάν αυτή η παράδοση νομολογίας την οποία αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τη μεταρρύθμιση, σε ποιο βαθμό λοιπόν αυτή η τήρηση θεμελιών δικαιωμάτων έχει επιπτώσεις και στις προβλέψεις των κρατών μελών. Ένα άλλο θέμα είναι η φροντίδα για τα άτομα που ε, έχουν ανάγκη από φροντίδες, που δεν αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά μόνο σε ορισμένα. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν τώρα προτείνει την ιδέα ότι η φροντίδα αυτή πρέπει να συμπεριληφθεί στο σύστημα συντονισμού των κοινωνικών παροχών. Δηλαδή, αυτά τα οποία έχει αναφέρει εδώ και δεκαετίες στην ε, νομολογία του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρέπει να ληφθούν υπόψη στη νέα αυτή ρύθμιση. Δηλαδή, η φροντίδα πρέπει να βασίζεται στις ε, βασικές αρχές ε, της ασφάλισης ασθενείας και πρέπει να μπορούν να εξαχθούν και εάν, εάν παρέχεται τέτοια φροντίδα πρέπει να γίνονται αποζημιώσεις των εξόδων με βάση τους βασικούς κανόνες συντονισμού. Αυτό που προκαλεί κάποιους εκνευρισμούς είναι ότι υπάρχει μια ρυθμίση που θέλει να εμποδίσει ότι οι παροχές φροντίδας και οι παροχές περίθλιψης ασθενείας πρέπει να εξετάζονται μαζί. Ο συντονισμός λοιπόν φτάνει σε κάποια όρια όταν ε, υπάρχουν ε, μεγάλες διαφορετικές διαφορές μεταξύ των κρατών που πρέπει να συντονίσουν την πολιτική τους. Μεγάλες διαφορετικές διαφορές, για παράδειγμα, θεωρείται η φροντίδα ως τμήμα της ε, παροχής υπηρεσιών περίθαλψης ασθενείας ή αν είναι χωριστό τμήμα. Στα διάφορα συστήματα λοιπόν κοινωνικής ασφάλισης η φροντίδα χρηματοοικονομικά και διοικητικά αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το σημαντικό τμήμα, κατά τη γνώμη μου, είναι η νέα διαμόρφωση των επιδομάτων και παροχών ανεργίας. Τι διαπιστώνουμε εδώ. Το ισχύον δίκαιο όσον αφορά τον συντονισμό των επιδομάτων ανεργίας ε, αποκλίνει κατά πολύ από, από τα άλλα τμήματα των κοινωνικών παροχών. Δηλαδή Μόνο περιορισμένα ισχύει η εξαγωγή των δικαιωμάτων ανεργίας. Ε, λαμβάνεται υπόψη ο συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης, αλλά υπάρχουν περιορισμοί για άτομα τα οποία κατοικούν σε μια χώρα και εργάζονται σε μια άλλη. Η πρόταση της Κομισιόν είναι αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς ε, να απαλληφθεί σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, οι παροχές ε, σε ε, επιδόματα ανεργίας, ε, οικονομικά ποσά, να είναι εγκυμένα για έξι μήνες και όχι μόνο για τρεις και κάτι άλλο, αναδιαμόρφωση της κοινωνικής κατάστασης και της κοινωνικής ασφάλισης των μεθοριακών εργαζομένων. Αυτό αφορά άτομα που εργάζονται σε μία χώρα ενώ ζουν σε άλλη. Στο μέλλον θα μπορούν να λαμβάνουν τα επιδόματα αυτά από το κράτος απασχόλησης. Δηλαδή θα υπάρξει ένα συντονισμό μεταξύ της χρηματοδότησης και του δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό ε, είναι πολύ θετικό κατά τη γνώμη μου. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τώρα οι κανόνε, όπου δεν ισχύει αυτή η αρχή, επειδή τώρα δεν ισχύει αυτή η αρχή, έχουμε μεγάλες δυσχέρειες. Δηλαδή για τον υπολογισμό των επιδομάτων, δηλαδή το τι ε, συνεισφορές πρέπει να έχουν ε, γίνει για να υπάρξουν κάποια επιδόματα, είναι πολύ ε, διαφορετικό για παράδειγμα στη Γερμανία από ό,τι στην Ελβετία. Από αυτά που δικαιούνται με βάση την χώρα διαμονής. Για παράδειγμα στην Ελβετία είναι πολύ ψηλότερο το επίπεδο των αποδοχών. Οπότε η αρχή είναι να είναι συγκρίσιμα τα επιδόματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και στη μία χώρα και στην άλλη. Με τον νέο κανονισμό θα σταματήσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή η αρχή της εξαγωγής των, ε, ε, παροχών θα έχει μεγάλα πλεονεκτήματα. Και ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι με βάση το ισχύον δίκαιο υπάρχει ανισορροπία μεταξύ του ότι το ότι κάποιος ο οποίος εργάζεται σε μία χώρα ε, πληρώνει φόρους σε αυτή τη χώρα αλλά τις παροχές τις παίρνει στη χώρα ορισμένες παροχές τις παίρνει στη χώρα διαμονής Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια εξισορρόπηση. Αυτός ο κανονισμός, όπως ισχύει μέχρι τώρα, δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί. Θα σταματήσει τώρα, εάν αλλάξουμε το σύστημα για τους ανέργους. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Αυτό όμως που θεωρώ ότι είναι προβληματικό είναι ότι οι βασικοί κανόνες των κρατών δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν για εργαζόμενους που θα έχουν εργαστεί για λιγότερο από 12 μήνες. Δηλαδή θα εξακολουθήσει να είναι το κράτος διαμονής υπεύθυνο για την παροχή αυτών των ε, επιδομάτων. Αυτό θεωρώ ότι είναι προβληματικό. Γιατί όποιος εργαστεί για μικρό χρονικό διάστημα δεν έχει δικαίωμα σε επιδόματα ανεργίας. Και τα συστήματα θα είναι πολύ διαφορετικά και περίπλοκα, άρα είναι δύσκολο να απολαύσει κανείς αυτά τα δικαιώματα. Και Τέτοιες καταστάσεις στην ουσία και για συγκεκριμένους σκοπούς, τους οποίους δεν θέλω να κακολογήσω, ε, τελικά προτιμούν ε, ιδιωτικές συμφωνίες εργαζόμενων τους εργοδότες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες αυτές και για την προσπάθεια σύνοψης αυτών. Δεν είναι κάτι εύκολο το λόγο στην κυρία Λιντογιόν. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα να σας μιλήσω για την νέα πρόταση κειμένου για τον κανονισμό που αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Βλίντε Γιόγκ. Ε, είμαι μέλος ενός διεθνούς δικτύου κοινωνικής ασφάλισης ε, και η συμμετοχή μου σήμερα στη συζήτηση θα αφορά πρακτικά ζητήματα. Τα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν υπάλληλοι και εργοδότες ε, όταν εργάζονται σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκα εγώ να συμμετέχω στη συζήτηση σήμερα. Έχω και μία παρουσίαση Κοιτώντας το κείμενο και την πρόταση κειμένου, θα περιοριστώ στο παροχές ενεργείας και αργότερα στη μακροχρόνια φροντίδα, κοιτώντας ε, τα επιδόματα ενεργείας και το προτινόμενο κείμενο, όπως είπε ο συνάδελφος, στην αρχή φαίνονται λογικέ ε, οι προτινόμενε αλλαγέ. Ουσιαστικά για του συνοριακού εργαζομένου, ε, το κράτο όπου εργάζονταν τελευταίο όπου ε, κατέβαλαν ε, συνεισφορές ε, κοινωνικής ασφάλισης θα είναι και το κράτος που θα πρέπει να καταβάλει τα επιδόματα ενεργείας το οποίο αν το συζητήσει κανεί με τις διασυνορικέ κοινότητε, θα το θεωρήσουν λογικό, διότι αυτή τη στιγμή κανονικά, αν είναι άνεργοι, το επίδομα ανεργία το πληρώνει το κράτο διαμονής, το οποίο είναι μια κάπως περίεργη κατάσταση. Φυσικά η αλλαγή στο κράτο τελευταία δραστηριότητα θα είναι πιο ενδιαφέρον σε περίπτωση εκεί το όταν το επιδομαριά είναι υψηλότερο. Ε, και φυσικά υπάρχουν άλλοι για του οποίου είναι πιο ευνοϊκή η σημερινή κατάσταση. Η μεταβολή αυτή στο τελευταίο κράτο απασχόλησης, το οποίο θα είναι αυτό που θα καταβάλει το επίδομα έχει και νόημα όσον αφορά τον εργοδότη, όταν κάνει ένα κοινωνικό σχέδιο ε, έτσι θα υπάρχει κάποια συνοχή ε, ε, ε, σε περίπτωση διασυνοριακού εργαζομένου θα πηγαίνει με το πλάνο της χώρας όπου εργάστηκε αντί για τη χώρα στην οποία κατοικεί. Και αν δει κανείς τις συνθήκες λήψης του επιδόματος ανεργίας, συχνά αν στο κράτος τελευταίας απασχόλησης για παράδειγμα ο υπάλληλο είχε συμφωνήσει με την απόλυσή του, ίσως το κράτο κατοικία του να του πει τότε δεν έχετε δικαίωμα για επίδομα ότι συμφωνήσατε να απολυθείτε. Οπότε υπάρχουν κάποια ωφέλη ε, στην προτινόμενη αυτή αλλαγή. Ε, πιστεύω θα πρέπει να το κοιτάξουμε πιο στενά. Ποια θα είναι ακριβώ ε, η επίπτωση της αλλαγή αυτής. Υπάρχουν μεταβατικοί κανόνες, ε, οποίους θα εισάγουν, ε, οι οποίοι θα εισαχθούν και πρέπει να δούμε κατά πόσο λειτουργούν πάντα σωστά ανάλογα με την κατάσταση. Επίσης ο συνυπολογισμός ε, της περίοδου 12 μηνών ε, για την οποία θα πρέπει κάποιος να έχει απασχοληθεί για 12 μήνες δηλαδή. Πώς θα υπολογίζεται αυτό 12 διαδοχικοί μήνες ή θα μπορούσε να είναι σπαστή ε, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πώς ακριβώς θα λειτουργεί και ε, σε ποιο σκεπτικό θα βασίζεται. Και επίσης ε, η υλοποίηση είναι κάτι που χρειάζει εξέταση. Η διασυνοριακή κοινότητα μπορεί ε, ένα διασυνοριακά εργαζόμενο θα έχει το δικαίωμα να αναζητήσει εργασία στη χώρα διαμονή του, ενώ θα λαμβάνει επίδομα από την άλλη χώρα στην οποία εργαζόταν τελευταία και πώς ε, ακριβώς θα οργανώνεται η καταβολή των επιδομάτων ενέργειας σε αυτή την περίπτωση. Κοιτώντα ε, ένα τώρα άλλο θέμα, ε, ένα νέο κεφάλαιο για τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας. Με πρώτη ματιά φαίνεται πολύ λογικό σαν να αποτελεί ουσιαστικά συνέχιση των όσων υπάρχουν ήδη ουσιαστικά εισάγεται ένα νέο κεφάλαιο το οποίο ε, μεταφέρει τους ίδιους σημερινούς κανόνες ε, ε, υγειονομικής περιθάλψης αλλά μα το δούμε από πιο κοντά βλέπουμε ότι η σημερινή διατύπωση θα οδηγήσει σε αλλαγή του συντονισμού των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ότι ορισμένοι άνθρωποι θα χάσουν παροχές όπως συνταξιούχοι που θα χάσουν κάποιες συντάξεις το οποίο θεωρούμε δεν ήταν ε, το σκεπτικό των προτινόμενων αλλαγών και επίσης θα είναι και πιο γραφειοκρατικό τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους οργανισμούς που θα εμπλέκονται σε αυτό. Εγώ αυτό που βλέπω επίσης είναι και το τι θα γίνεται στην καθημερινότητα και πιστεύω ότι σας απασχολεί και εσάς. Πώς το βλέπουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Όταν τους μιλώ μου λένε ότι η σημερινή πρόταση για αυτούς δεν αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα τα πράγματα έτσι όπως έχουν σήμερα. Αυτό που λέω το πιο δύσκολο ε, με τους ε, διεθνείς εργαζομένους θα είναι να μπορούμε να παρακολουθούμε πού βρίσκεται ο καθένας, ε, πώς θα συμμορφωθούμε με τους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης, και τι γίνεται όταν κάποιο ε, τεθεί υπό το σύστημα κοινωνική ασφάλιση μια άλλη χώρα. Κάτι πολύ πιθανό σε έναν κόσμο που ο κόσμο κινείται περισσότερο, επιτρέπεται να εργαστεί από το σπίτι του. Και εκεί το σύστημα κοινωνική ασφάλιση μπορεί να είναι αυτό τη χώρα κατοικία και συχνά ένα εργοδότη έχει να αντιμετωπίσει και να εγγράψει τον υπάλληλο στην χώρα διαμονή του, ε, να συζητήσει με ε, αρχέ ξένων χωρών. Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλο φόρτο τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο. Συζητώντας με τους διαφορούς ενδιαφερομένους, έμαθα ότι η εισαγωγή ενός μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ενιαίας στηρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μπορούσε θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα ε, που θα βοηθούσε την ελεύθερη μετακίνηση για οποιονδήποτε θέλει να τεθεί στο ε, σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μια άλλη χώρα. Επίση, τώρα κοιτώντα ε, και τον μεταβαλλόμενο κόσμο μα υπάρχουν διάφοροι καινοτόμοι τρόποι εργασία, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον. Όταν σχεδιάστηκε στην αρχή ο κανονισμό, το να εργάζεται κανεί διεθνώ ή από το σπίτι του δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο, αλλά σήμερα πολλοί εργοδότες δίνουν κίνητρα στους υπαλλήλους τους να μην εργάζονται στο γραφείο, αλλά στο σπίτι, σε ένα γραφείο ενδεχομένω εντό τη οικία του. και δεν κάνουν τη διαφορά μεταξύ εθνικών εντό εισαγωγικών εργαζομένων και διεθνών, φυσικά. Είναι κάτι που δεν επιτρέπεται. Αλλά αν κάποιο ε, διασυνοριακό εργαζόμενο μπορεί να εργαστεί από το σπίτι του, αυτό σημαίνει ότι επειδή εργάζεται από το σπίτι του, η κοινωνική του ασφάλιση θα πρέπει να αλλάξει. Ε, όπως ξέρετε, αν εργάζεται κανείς 20, κατά 25% στη χώρα κατοικίας του, θα πρέπει να υπόκειται στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσης της χώρας ε, διαμονής του. Και δεδομένου των σύγχρονων μορφών εργασίας αυτών λοιπόν, που είπαμε, αυτό θα δημιουργήσει διαφορές ε, ε, μεταξύ της διεθνούς και της εθνικής της διεθνούς και του εθνικού εργατικού δυναμικού. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν κατά πόσο οι κανόνες συντονισμού μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο. Από την ίδια άποψη, κοιτώντα τους κανόνες συντονισμού για τους απεσπασμένους εργαζομένους και για την εργασία σε πολλά κράτη, όταν συντάχθηκε ο κανονισμός στην αρχή πριν πολλά πολλά χρόνια, ένα απεσπασμένο εργαζόμενο ήταν κάποιος που μετέβαινε σε μια άλλη χώρα και δούλευε εκεί 100% του χρόνου του αλλά σήμερα ο κόσμος έχει γίνει πολύ μικρότερος, ο κόσμος κινείται πιο εύκολα και συχνά μια διεθνή αποστολή σημαίνει ότι η απόσπαση σημαίνει ότι κάποιο πρέπει να εργάζεται σε πολλέ ερωτικέ χώρε ή να επιστρέφει καμιά φορά στη χώρα από την οποία σταλεί. Έτσι με τους σημερινούς ε, κανόνες δεν μιλάμε για απόσπαση αλλά για εργασία σε πολλαπλά κράτη το οποίο σημαίνει ότι αν κάποιος μεταφέρει ε, την διαμονή του στη χώρα απόσπασή του θα πρέπει να αλλάξει και σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ε, κάτι ανεπιθύμητο τόσο από τον εργαζόμενο όσο και τον εργοδότη. Οπότε οι συμφωνίε σε δυνάμει του 16 μπορούν να συναυτούν αλλά είναι πολύ ε, σκηνοτενεί διαδικασίε. Ε, πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν εκτενέστερα, μήπω πρέπει να αλλάξουν οι κανόνε γι' αυτό. Έχω και το παράρτημα, το οποίο μπορώ να σας ε, δώσω αργότερα και το οποίο περιλαμβάνει διάφορα άλλα θέματα, το οποίο πιστεύω αξίζει να εξετάσουμε. Είναι πολύ τεχνική φύση, πολύ αναλυτικά, οπότε θα τα αφήσω για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας και ιδιαίτερα για το πώ θέσατε το θέμα των ε, υπέρ και τα κατά και για τους εργοδότες και για του εργαζόμενου, και ιδιαίτερα το θέμα των νέων επαγγελμάτων που και αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αντιμετώπιση μας και νομίζω ότι έχουμε εδώ και μια ομάδα επισκεπτών της κυρίας Μογάν Σάτχε από ένα λύκειο πρότυπο καινοτόμο και διεθνές του Πουατιέ που είναι μια γαλλική πόλη που την γνωρίζουμε ακριβώς για το ότι είναι, για το ότι είναι κέντρο καινοτομίας και είναι ιδιαίτερα στραμμένη προς το μέλλον. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίασή μας. Και τώρα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Κάρλος Καρθία Δεκορτάθαρ Νεβράδα. Δέκα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη συνεδρίαση αυτή. Εγώ, αν ήμουν νομοθέτης ή ε, συνεγράφα βιβλία για τα θέματα αυτά, θα έβαζα ως υπότιλο στα, γραφεία, στα βιβλία μου αυτά για την ε, ε, κοινωνική ασφάλιση που θα έλεγε ότι αν το διαβάσετε χωρίς ε, πρώτερη προετοιμασία μπορεί να έχετε σοβαρά προβλήματα υγείας. Τι εννοώ. Εννοώ ότι διαβάζοντας ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματικά μπορεί να έχει βλαβερές συνέπειες. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει τόσο σοβαρές συνέπειες. Δεν θα υποφέρεται πολύ. Όταν πρώτο διάβασα τον κανονισμό 1408 προετοίμαζα την ένταξη της Ισπανίας ε, της Ένωσης και είπα στον εαυτό μου Κάρλος δεν καταλαβαίνεις μία, είσαι ανόητος. Σιγά σιγά κάτι άρχισα να καταλαβαίνω. Άρα μην απελπίζεστε. Εάν ορισμένα από αυτά που λέει η πρόταση δεν τα καταλαβαίνετε. Ο κανονισμός 883 ξεκίνησε το 1996 και τελικά εγκρίθηκε το 2004. 7 χρόνια διαπραγματεύσεων κατόπιν άρχισε να ισχύει το 2010. Δηλαδή 13 χρόνια από την παρουσίαση από πλευράς της Κομισιόν του αρχικού σχεδίου. Άρα πρέπει να καταλάβετε ότι οποιαδήποτε τροποποίηση σε αυτή την τόσο περίπλοκη νομοθεσία δύσκολα θα επιτευχθεί με βάση συνένεση. Γιατί η πρόταση της Κομισιόν αντιμετωπίζει ε, πολύ διαφορετικά τμήματα, πολύ διαφορετικές ε, πλευρές αυτού του κανονισμού. Αλλά στην ουσία ένα είναι το κύριο. Η καταπολέμηση των ε, απατών, κατά των καταχρήσεων. Το θέμα όμως είναι ότι καταπολεμώντας τις απάτες και τις καταχρήσεις, επί, των οποίων, επί της οποίας όλοι συμφωνούμε, πρέπει να δούμε αν τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι τα ανάλογα. Από τότε που εγκρίθηκε ο κανονισμός 883 έγινε μόνο μια πολύ μικρή έκταση τροποποίησή του το 2010. Αλλά η πρόταση αυτή θα έλεγα ότι είναι πολύ σχηδής γιατί αντιμετωπίζει πολλές πλευρές. Πρέπει να την εξετάσουμε αναλυτικά και θα σας ε, υποβάλω δύο ιδέες. Σε αυτή την πρόταση υπάρχουν ε, στοιχεία καθαρά πολιτικά και στοιχεία καθαρά τεχνικά. Μεταξύ αυτών των πολιτικών και τεχνικών ε, στοιχείων θα αναφερθώ σε τρία θέματα. Ορισμένα τα ανέφεραν ήδη οι προηγούμενοι ομιλητέ. Και επαφίεμαι σε εκείνου, γιατί οι παρουσιάσει του ε, ήταν πολύ σωστέ. Ίσως να προσθέσω κάτι ακόμη. Το βασικό είναι, είναι η αρχή ίσης μεταχείρισης. Έχουμε την ιδεολογική σκέψη 5 που είναι στοιχείο κλειδί για να καταλάβουμε την πρόταση. Και ιδιαίτερα για να καταλάβουμε το άρθρο 4 παράγραφος 2. Εδώ αναφερόμεθα στην αρχή ίσης μεταχείρισης. Αλλά υπό προϋποθέσεις. τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, εισαγάγουν περιορισμούς για τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης για τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες. Ωραία. Αυτή είναι μια διατύπωση που βασίζεται στην ομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αλλά ακριβώς από την ομολογία, όχι ακριβώς. Ας πούμε ότι πάει ακόμη παραπέρα. Αντίθετα με το δικαστήριο, το οποίο θέτει ορισμένες κόκκινε γραμμές, η πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής τις υπερβαίνει. Και να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί το λέω αυτό. Ορίστε, δείτε μία υπόθεση εδώ. Μία από τις πιο σημαντικές υποθέσεις ε, επί των οποίων βασίστηκε η πρόταση της Επιτροπής. Είναι η υπόθεση Pizza Bray. Τι λέει το δικαστήριο για αυτή την υπόθεση ότι δεν είναι δυνατόν να καταργείται αυτόματα η ισότιμη μεταχείριση υπό ιεσδήποτε συνθήκες. Αν διαβάσουμε συγκεκριμένα ή διαφορετικά, θα ερμηνεύσουμε ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες υπό τις οποίες δεν υπάρχει αυτός ο αυτοματισμός. Ας πάρουμε τώρα την πρόταση. Ας την ερμηνεύσουμε. Ορισμένοι την ερμήνευσαν αλλά δεν ανταποκρίνεται βέβαια κυριολεκτικά σε αυτά που λέει η πρόταση. Γιατί θα είναι σαν να δίνουμε ελευκό επιταγή, ούτω ώστε ορισμένε χώρε να εξαιρούν μια σειρά από εξαιρέσει. Να μην παρέχουν λοιπόν αυτές τις ε, παροχές σε κάποια μη οικονομικά ενεργά άτομα. Δηλαδή ανοίγουμε το κουτί της πανδώρας. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι αυτό λέει νομολογία. Ναι, σε ορισμένε περιπτώσει. Στην περίπτωση του Peter Bray, που είναι πολύ σημαντική υπόθεση, σχετικά πολύ σημαντική, γιατί υπήρξε και, και μία αγωγή του, ε, της Επιτροπής κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Και η Επιτροπή, ε, συγγνώμη, το δικαστήριο ε, απεφάνθη υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν πριν από τον Brexit. Θα αναφερθώ όμως ορισμένα στοιχεία αυτής της απόφασης. Το δικαστήριο αποδέχεται ότι υπήρξε έμεση διακριτική μεταχείριση. Δεύτερον, το δικαστήριο θεωρεί ότι αυτή η έμεση διακριτική μεταχείριση μπορεί να έχει επιπτώσεις ε, στους πόρους του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά κυρίως απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής, κυρίως γιατί λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, παρήχε επαρκή στοιχεία και αιτιολόγηση. Και τι σημαίνει αυτό. Εάν στο μέλλον η Κομισιόν ε, υποβάλει επαρκή αιτιολόγηση, τι θα γίνει. Τότε θα μπορούσε να έχει υπάρξει άλλη απόφαση που να είναι αντίθετη λοιπόν στην αρχή της ισότιμη μεταχείρισης. Ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται αυτή η απόφαση, συγγνώμη, μάλλον αυτή η πρόταση κανονισμού, σημαίνει ότι αποδεχόμεθα κάτι που ούτε καν το δικαστήριο δεν είχε ποτέ ορίσει. Εσείς θα το αποφασίζετε αυτό, όχι εμείς. Εάν θα εγκρίνετε δηλαδή την πρόταση. Αλλά με την πρόταση αυτή πρέπει να πω ότι φτάνουμε στα όρια της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Και αυτό είναι βασικό, μάλλον των ε, ατόμων. Και δεν θα μιλήσω τώρα για τα επιδόματα ανεργίας, γιατί οι προηγούμενοι ομιλητές ε, είπαν πολλά και συμφωνώ απόλυτα αλλά να κάνω μία ε, μικρή αναφορά σε ορισμένα. Για πρώτη φορά στο κείμενο αυτό, σε κανονισμό δηλαδή, προβλέπεται μία περίοδος αναμονής τριών μηνών. Δηλαδή, κάποιο κράτος πρέπει να αποφασίσει για το πότε θα κάνει αυτές τις παροχές. Και γίνεται συνυπολογισμός και των συνεισφορών σε προηγούμενο κράτος. Αλλά εάν στο τελευταίο κράτος που συνεισφέρει στην κοινωνική ασφάλιση δεν έχει συνεισφέρει για τρει μήνες, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να έχει επιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις. Τι θα μπορούσε να συμβεί. Ένα άτομο. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Ένας εργαζόμενος που έχει εργαστεί 24 ε, μήνες σε ένα κράτος και μετά πάει σε ένα άλλο κράτος. Εργάζεται δύο μήνες και μετά χάνει τη δουλειά του το δεύτερο κράτος θα έπρεπε να του χορηγήσει επιδόματα ανεργίας συνυπολογίζοντα την περίοδο που έχει εργαστεί και στον προηγούμενο κράτο. 24 συν 2, 24 συν 2, 26 μήνε. Με την πρόταση τη Κομισιόν, όπου έχει εργαστεί 24 στο κράτο Α και μετά, ε, ε μετά αλλάζει ε, τον τόπο εργασία στο κράτο Β, εάν μετά μείνει άνεργο το άτομο αυτό, θα πρέπει το κράτο Α να του δώσει τα επιδόματα ανεργία. αλλά δεν δηλαδή, έχει καμία σχέση πλέον με το κράτο Α εφόσον, παραμένει, εφόσον διαμένει στο κράτος ε, Β. Και μπορεί να είναι ε, οι παροχές που θα πάρει από το κράτος Α, ανεπαρκής για το επίπεδο ε, το βιωτικό, το επίπεδο αποδοχών του κράτους Β και μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερες. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με το άρθρο 48 που λέει ότι πρέπει να συνυπολογίζονται όλες οι περίοδοι. 48 τις συνθήκες Όλες οι περίοδοι. Εδώ εισάγεται μία μικρή τροποποίηση στην ερμηνεία του άρθρου 42 και καταλήγω. Υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο. Εκτελεστικές πράξεις και κατεξοδότηση πράξεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά τις σχέσεις ε, των τριών θεσμικών οργάνων. Να σας πω ότι αν μου θέσετε την ερώτηση, ποια είναι η γνώμη μου, αλλά θα σας αφήσω εσάς να με ρωτήσετε. Κάτι που κάνατε το 2009-10 όταν τροποποιήσατε ένα παράρτημα θα σας το εξηγήσω. Τώρα δεν θα μπορείτε να το κάνετε. Κάτι το οποίο επιτύχατε ούτω ώστε τα μέλη της οικογένειας των διαμεθοριακών εργαζομένων να έχουν κάποια δικαιώματα δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να το κάνετε. Και μπορώ να σας δώσω πολλά άλλα παραδείγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την ενημέρωση μας προκαλεί διαφορε σκέψεις και φυσικά θα μα δίνει να σκεφτούμε ότι πρέπει να σκεφτούμε και πώ θα προχωρήσουμε και όσον αφορά την απόφαση του δικαστηρίου. Δίνουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μπαλά, στον εισηγητή μα για τρία λεπτά. Ναι, ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια αυτά τα οποία δεν δείχνουν τίποτα άλλο από το ότι είναι περίπλοκο το ζήτημα αυτό σήμερα η πρόθεση αυτή της Κομισιόν πρέπει πράγματι να ε, αναλυθεί από εμάς, ε, να, την, ε, να υποστεί επεξεργασία για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θα μιλήσω πολύ γιατί θέλω να αφήσω τον περισσότερο δυνατό χρόνο για ερωτήσεις στους όδης βέβαια αλλά και στο σύνολο των συναδέλφων μου. Ωστόσο ήθελα να ρωτήσω τον καθένα από τους ειδικού που ακούσαμε εδώ σήμερα γιατί ομολογώ ότι δεν περίμενα τέτοια είδους ανάλυση και τόσο μεγάλη απόσταση σε σχέση με τις προτάσεις της Κομισιόν. Πέραν λοιπόν των όσων εσείς επισημάνατε, ε, πολύ συγκεκριμένα, θα μπορούσατε να μου κάνετε μια πιο γενική εκτίμηση, αποτίμηση όλων των προτάσεων της ε, Κομισιόν σήμερα. Δηλαδή θεωρείτε ότι αυτές οι προτάσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και χρειάζεται να βελτιωθούν. Πιστεύετε ότι πρέπει να τις αλλάξουμε, να τις μεταρρυθμίσουμε και να τις βελτιώσουμε διότι αλλιώς θα περιπλέξουν υπερβολικά το σύνολο. Θέλω να μας μιλήσετε απολύτως ελεύθερα και να μας δώσετε τη γενική εντύπωση που έχετε σχηματίσει ε, μια πιο γενική εικόνα, ώστε να έχουμε μια συνολική εικόνα και εμείς. Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο τώρα στους διάφορους ε, σκιώδεις. Και στη συνέχεια οι τρεις, ε, εδώ, τα τρία μέλη του πάνελ θα μπορέσουν να απαντήσουν στις διάφορες ερωτήσεις που σίγουρα θα ακούσουμε ε, και που θα προσταθούν σε όσους ακούσαμε τώρα. Ε, δίνω λοιπόν δύο λεπτά σε κάθε σκιώδη για το ΕΛΚ ο κύριος Φένσης. Παρακαλώ. Αγαπητά κύριε Πρόεδρε, Καθηγητά Άχενχόφερ, κυρία Ντεγιόν, κυρία Κρασία, σας ευχαριστώ πολύ καταρχάς που ήρθατε. Θα πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα η τελευταία παρουσίαση μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, διάβασα την νομοθεσία, πολλές σελίδες, το πώς μπορούμε να την ερμηνεύσουμε, όπως είπατε και εσείς. Πιστεύω όμως πως η βάση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετά καλή. Ήθελα όμως να κάνω και μερικές ερωτήσεις. Θα είμαι σύντομος λοιπόν, γιατί αναφερθήκατε ήδη σε ορισμένες από αυτές. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξηθεί ο χρόνος ε, του επιδόματος ενεργής από 3 σε έξι μήνες, ακούσαμε ότι είναι έτσι, μια καινούργια πρόταση. Εσείς, κυρία καθηγητά Άχενχοφερ, θεωρείτε πως είναι σωστό αυτό το χρονικό διάστημα, είναι αρκετό. Επίσης, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αναθεώρηση του κανονισμού 883. Εσείς θεωρείτε πως έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό. Μετά, να αναφερθώ στην υπόθεση Αλεμάνοβιτς, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ε, νομοθεσία αυτή αποκλεί λοιπόν τον δικαιούχο από την ε, έλλειψη αυτών των επιδομάτων. Εσείς θεωρείτε σωστή αυτή την απόφαση. Ε, αυτά για τα δύο λεπτά που έχω χρόνο. Αν καταφέρω μετά θα ε, σας κάνω και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δίνω το λόγο στην κυρία Χέλγκα Στίβενς. Thank you, Chair. Oh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Η μία είναι όμοια με αυτή του συναδέλφου μου ε, για το πώς δηλαδή μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πώς μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε στην πρόταση. Η πρόταση συμπεριέλαβε κάποιες από τις αποφάσεις του δικαστηρίου Και θεωρώ πως η πρόταση παρέχει πολύ χρήσιμες διευκρινήσεις και θα μας δώσει έτσι περισσότερη ασφάλεια δικαίου. Και για τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορούν να καθορίσουν τι ε, χρειάζεται έτσι ώστε να αποδείξει ένα άτομο ε, τη διαμονή του εκεί και να μπορεί να λάβει αυτές τις παροχές. Έχω καταλάβει σωστά. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Τώρα, να περάσουμε και στην εξογή των ε, παροχών για τα παιδιά. Έχω αναφερθεί στο θέμα αυτό στο παρελθόν ε, και θεωρώ πως συνεχίζει να είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει προσπάθεια να ε, μειωθούν στο ελάχιστο αυτές οι εξαγωγές των επιδομάτων για τα παιδιά. Πώς μπορούμε όμως να αντιμετωπίζουμε το κάθε παιδί με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν πολλές διαφορές στην Ευρώπη, πολλές ανισότητες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και αν κατάλαβα καλά, η Επίτροπος Τάισεν είπε στην ακρόαση ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό, 1 ή 2% το πολύ, αυτών που χρησιμοποιούν αυτές τις ε, διατάξεις για να λαμβάνουν επιδόματα παιδιών. Αλλά για κάποιες άλλες χώρες είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Σίγουρα, ένδουμε το μέσο όρο σε όλη την επικράτεια της Ένωσης, είναι πολύ χαμηλός, όμως υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία έχουν πολύ ψηλότερα ποσοστά και μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό θα ήθελα να δούμε ε, πιο λεπτομερώς το θέμα αυτό. τώρα, ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης της απάτης ή της κατάχρησης του συστήματος. Αυτό που βλέπω είναι πως τα κράτη-μέλη ε, χρειάζονται έναν ενιαίο ε, τρόπο, ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης αυτών των περιπτώσεων. Εσείς θεωρείτε πως ε, έχει δείξει αποτελέσματα μέχρι τώρα αυτό το σύστημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρία Νάκιν για την ομάδα Άλτε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους εμπειρογνώμονες. Σίγουρα το κείμενο είναι πολύπλοκο και έχουμε όλοι πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχω όμως κάποια σύντομα σχόλια οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου νομίζω ελήφθησαν με μεγάλη ε, προσοχή. Ήταν προσεκτικές. Ο τελευταίος ο αναφέρθηκε σε αυτές και αναφερθήκατε επίσης στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρήχε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη μετακίνηση των ε, Ατόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ε, ποια είναι, ποιες είναι οι δυσκολίες που εντοπίζουμε εδώ. Όταν διαβάζω εγώ μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν μπορώ να την ερμηνεύσω με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Η απόφαση είναι μια απόφαση. Θα ήθελα λοιπόν τα σχολιά σας πάνω σε αυτό. Και ε, προς την κυρία Ντεγιόμ. Αναφερθήκατε στο πώς μπορεί ένα κράτος μέλος να διασφαλίσει πω ένας άνεργος πληρεί όλες τι αναγκαίε προποθέσει ώστε να λάβει πληρει ολες τις αναγκαιε ανεργίας. λαβει επιδομα ενεργειας διορθωστε με αν κάνω λάθος, αλλά προτείνετε δηλαδή εσείς ότι όταν κάποιος πηγαίνει από τη χώρα Α στη χώρα Β και στη χώρα Β έχει πρόσβαση σε επιδόματα ενεργείας από τη χώρα Α αυτό δεν είναι το ίδιο με ένα, με ένα άτομο οποίο, το οποίο έχει παραμείνει στη χώρα Α και λαμβάνει επιδόματα εκεί. Μας είπατε επίσης ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τους εργοδότες είναι η γραφειοκρατία, ε, διοικητική και τα, η μεταφορά ε, ε, επιδομάτων από τη μία χώρα στην άλλη. Κατάλαβα τι εννοείτε. Δεν είμαι σίγουρη όμως πόσο σχετικό είναι με αυτό που συζητάμε και με τις επιπτώσεις στην νομοθεσία. Τώρα έχω άλλες 10 ερωτήσεις, ίσως και 100 ερωτήσεις που θα μπορούσα να κάνω, δεν ξέρω όμως αν θα έπρεπε. Έκανα όμως την αρχή. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε με τις πρώτες ερωτήσεις, αλλά ναι, φυσικά θα ακολουθήσουν πολλές άλλες ε, κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Για δύο λεπτά τώρα, η κυρία Τσιμέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πυρογνώμονες. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ με τις παρουσιάσεις σας και νομίζω πως θα ήταν πολύ καλό για μας να τις είχαμε και γραπτός. Τώρα, ας έρθω στο θέμα. Ελάχιστη διάρκεια εξαγωγής των ε, παροχών. Μας ε, είπατε πως υπάρχει πρόταση να αυξηθεί το διάστημα από τους τρεις στους έξι μήνες. Αλλά από αυτά που άκουσα μου φαίνεται πως ε, θέλετε λιγότερη γραφειοκρατία για όσους αναζητούν εργασία στα πλαίσια της ελεύθερης μετακίνησης και πως ε, αυτό είναι καλό να γίνει με την νέα νομοθεσία. Επίσης μιλήσατε για το, την ανάγκη να μην περιοριζόμαστε στους 12 ε, μήνες απασχόλησης. Δεν έχω καταλάβει όμως ε, τα επιχειρήματα υπέρ και κατά για να είμαι ειλικρινής. Μετά, οι διατάξει σχετικά με το δικαίωμα διαμονής. Πώς αυτό ε, μπορεί να συνδεθεί με την, το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης. Εδώ θα ήθελα να μάθω τις δικές σας εκτιμήσεις για την πρόταση της Επιτροπής, βασισμένη όμως στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τις αποφάσεις που αφορούν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης όλων των πολιτών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εάν αυτές, αυτή η ελεύθερη μετακίνηση αφορά και τη μετακίνηση των εργαζόμενων. Και μετά υπάρχει και το πρόβλημα των αστέγων. Εσείς βλέπετε κάποια άμεση συσχέτιση με την πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι άστεγοι που έχουν μεταβεί σε άλλη χώρα, οι οποίοι ήδη έχουν προβλήματα πρόσβασης σε κοινωνικές παροχές. Νομίζετε πως θα αυξηθεί ο ρυθμός των αστέγων. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την κυρία Ατζία για το EFDD. Υπάρχει κανείς για να την αντικαταστήσει. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Κυρία Λάμπερτ, σας ξέχασα. Να σας δώσω το λόγο. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Βεβαίως ε, με ενδιαφέρει πολύ το θέμα αυτό. Έχω εμπλακεί, ήμουν εισηγήτρια για τον κανονισμό 883 και για τον εφαρμοστικό του κανονισμό. Συγγνώμη, συγγνώμη για τα κενά που έχουν τα κείμενα αυτά, αλλά χρειαζόταν ομοφωνία στο Συμβούλιο, αλλά δεν μπορούσα να κάνει και πολλά το Κοινοβούλιο. Να αναφερθώ σε ορισμένα που υπόθηκαν. Πρώτον, για το άρθρο 4 παράγραφος 2, το θέμα της ε, ίσης μεταχείρισης. πρόταση που έχει υποβληθεί στην ουσία είναι πισωγύρισμα. Μειώνεται η συμμεταχείριση. Και ανα, αναφερόμενοι σε μία συγκεκριμένη απόφαση του δικαστηρίου, αμφισβητούμε τα δικαιώματα ενός μεγάλου αριθμού πολιτών της Ένωσης. Πρώτα απ' όλα οι οικονομικά ανενεργοί είναι για παράδειγμα συνταξιούχοι είναι άτομα που μπορεί να χρειαστεί να φροντίζουν ε, τον οικοκυριό ενώ ο σύντροφός τους εργάζεται. Πολλοί μπορεί να έχουν παράγωγα δικαιώματα. Είναι σαφές αυτό που κάνουμε τώρα για τα άτομα με παράγωγα δικαιώματα. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε την αρχή της ίσης μεταχείρισης, γιατί θα προκύψουν πραγματικές δυσχέρειες. λόγω ακριβών αλλαγών στα δικαιώματα των ε, πολιτών της Ένωσης λόγω της απόφασης για τον Brexit. Τώρα για τις ε, σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας και το θέμα ότι πρέπει να εργαστείς στο κράτος ε, Β τρεις μήνες πριν να αποκτήσεις δικαίωμα σε ορισμένες παροχές εκεί. Πώς θα καθορίσουμε τι σημαίνει τρεις μήνες. Ορισμένοι αρχίζουν να εργάζονται στην αρχή με άτυπε μορφές εργασία, με μερική απασχόληση. Υπάρχουν πολλά τέτοια φαινόμενα. Πώς θα υπολογιστεί. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Επίσης θέσατε το θέμα για τους διαμεθοριακούς που μπορεί τελικά να θυγούν ή μάλλον θίγονται με τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Διαμεθοριακοί εργαζόμενοι, δηλαδή ζω στη μία χώρα, εργάζομαι στη διπλανή. Τι θα έπρεπε να κάνουμε για αυτούς. Και τέλος, τι ακριβώς ε, δεν ε, μπόρεσε να συμπεριλάβει η πρόταση που έχουμε τώρα ενώπιον μας, τι μπορούμε να προσθέσουμε για να διευκολύνουμε τα άτομα που ε, προσπαθούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε ελεύθερη κυκλοφορία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Ε, δεν βλέπω την κυρία Μίλων, ίσως ο κύριος Μαρτάν. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Κατάλαβα πολύ καλά τι είπε ο κύριος Γκαρθία Κατάλαβα τι είπε η κυρία Ντεγιόν, αλλά αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής Άχενχόφα, ίσως ε, δεν τα κατάλαβα καλά. Κοιτάξτε, εγώ ε, τώρα πρώτο κοιτάζω το κείμενο, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικών παροχών. Θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο για οικογενειακά επιδόματα, για ασφάλιση ασθενείες, ενώ μιλάμε μόνο για τα επιδόματα ανεργίας. Αυτό είναι η πρώτη μου έκπληξη. Κατάλαβα τους τρεις ομιλητές που είπαν ότι στόχος μας είναι να υπάρξει εναρμόνιση και σύγκληση. Α, ευσεβής πόθη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εδώ και χρόνια. Αλλά φοβάμαι ότι εξετάζουμε αντίστροφα τα πράγματα. θα έπρεπε νομίζω να έχουμε προωθήσει κάτι το οποίο είναι αντίθετο από αυτό που θέλετε. Πριν ευνοήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία, την κινητικότητα των εργαζομένων, την ε, ασφάλεια, την οδηγία για τους αποσπασμένους, πρώτα θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την εναρμόνιση και σύγκληση της Ευρώπης των 6, των 7. Όχι να επιχειρούμε τώρα να κάνουμε λοιπόν τα πράγματα με λάθος σειρά είναι σαν το βάτροχο που ε, άρχισε να φουσκώνει, να φουσκώνει, να κρατάει την αναπνοή του για να γίνει μεγάλος σαν βόδι και έσκασε. Είναι αντιφάσεις αυτά τα πράγματα. Και καταλήγω με μια ε, πολύ απλή παρατήρηση. Δεν θεωρείτε ότι ο πιο εύκολος κανόνας ε, και ο πιο δίκαιος θα ήταν όποιος λαμβάνει τις συνεισφορές και των εργαζομένων και των λογοδοτών σε κάθε κράτος μέλος, όπου ακριβώ εργάζεται ο εργαζόμενος, αυτός θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τα επιδόματα. Γιατί τώρα να λέμε να τα αναλάβει η χώρα Α, η χώρα Β με προράτα, τέμπορις, με βάση το χρόνο εργασίας σε κάθε χώρα, όλα αυτά είναι πολύ περίπλοκα. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον εισηγητή και τους Σκιώδης. Να δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους μας ε, ε βουλευτές, η κυρία Μαρή Αρενά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις. Έχω την εντύπωση ότι στην πρόταση συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης όταν μιλάμε για την πρόσβαση σε παροχές οικογενειακές, ανεργίες κλπ. Υπάρχει μια αρχή περισσότερο περιορισμού, περιορισμού δηλαδή της ελεύθερης μετακίνησης, της ελεύθερης κυκλοφορίας. Αντιθέτως, ε, ε, το λιγότερο σαφές πράγμα είναι το, ε, στον κανονισμό αυτό είναι αυτό που αφορά την απόσπαση. Ε, φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα αντίστροφα όταν μιλάμε για καταπολέμηση της απάτης στο πρώτο κομμάτι με περιορισμό των πρόσβασης ακολουθείται αντίστροφη φιλοσοφία στο θέμα της απόσπασης εργαζομένων. Εγώ έχω μια πολύ σαφή ερώτηση για το πώς θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα πράγματα ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας από κοινού με ό,τι γίνεται με την οδηγία για την απόσπαση. Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου βάσει μιας πρότασης της Γερμανίας που είναι βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης. Δηλαδή η ε, επιχείρηση η οποία ε, έχει απασχολήσει τον εργαζόμενο μπορεί να ε, φυλάξει ως εχέγγιο τα ε, ποσά αυτά ώστε να παρασχεθούν αργότερα στην ε, επόμενη χώρα. Αυτό πρότεινε το δικαστήριο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει αυτή η αρχή στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης γιατί αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες περιπτώσεις απάτης. Ε, και λόγος για τον οποίο δεν ε, καταβάλλεται ένα επίδομα ενεργείας ε, από την αρχική χώρα. Το δεύτερο ζήτημα είναι η έκδοση του εγγράφου Α1 που είναι ένα σημαντικό εγγραφό το οποίο εγγυάται ότι υπήρξε εργασία στην αρχική χώρα όταν το στέλνουμε στη δεύτερη χώρα. Και θα μπορούσε αυτό να λειτουργεί σήμερα αναδρομικά, δηλαδή σε περίπτωση που υπάρξει έλεγχος και δεν υπάρχει, μπορεί να εκδοθεί το έγγραφο στη συνέχεια. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να λέμε ότι το έγγραφο αυτό θα, γίνεται, θα δίνεται προληπτικά, δηλαδή να λέμε ότι χρειάζονται τρεις μήνες τουλάχιστον εργασία στην αρχική χώρα και να δίνεται το α1. Αυτό όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Ή το τρίτο ερώτημα θα μπορούσε να υπάρχει ένα μητρό ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δηλαδή τι, ένα μητρό ενημέρωσης που θα μας λέει ποια είναι η κατάσταση των χωρών στη χώρα καταγωγής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο Βέλγιο, όταν κανείς δεν έχει πληρώσει τις κοινωνικές του εισφορές, έχει ένα κόκκινο αναγνωριστικό στην επιχείρηση όταν μια επιχείρηση έχει ένα τέτοιο κόκκινο αναγνωριστικό στο μητρό επιχειρήσεων, δεν έχει πρόσβαση στους, ε, στους πληστηριασμούς, ας πούμε, στις, ε, στους δημόσιους διαγωνισμούς. Ενώ σε άλλες χώρες μπορεί. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει ένα τέτοιο μητρό ευρωπαϊκό, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ όλων των επιχειρήσεων. Προβλέπετε κάτι τέτοιο ε, στο συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση. Ευχαριστούμε. Ζωσδακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν έχω καταλάβει καλά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόκειται καταρχάς για καλύτερη κοινωνική προστασία και για ε, περισσότερη δικαιοσύνη και για αποφυγή καταχρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπε και η κυρία Στίβενς ήδη, και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το ότι υπάρχει αυτό το 1 έως 2% περιπτώσεων κατάχρησης της νομοθεσίας. Αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι σε αυτό όπως είπα. Ε, αυτό που χρειάζεται είναι ενίσχυση των ελέγχων. Γι' αυτό διερωτώμε εάν εδώ θα έχουμε ένα πρόσθετο μεγάλο διοικητικό φόρτο. Χρειάζονται διμερείς συμφωνίες ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό έχω κάποιες επιφυλάξεις. Νομίζω πως στο μέλλον δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την κατάσταση, ούτε και να ανταποκριθούμε στον τεράστιο διοικητικό φόρτο που θα επιφέρει η αλλαγή της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντσαντέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ. Ε, είναι πολύ σημαντικό να... που κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και βλέπετε τελικά αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι μας έχουμε πολλές ερωτήσεις και θα έχουμε όλο και περισσότερες όσο θα προχωράνε οι εργασίες μας. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο αφορά την κατάσταση των ε, διαμεθοριακών εργαζομένων. Αναφέρθηκε ήδη. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια έχουμε δύο τύπους εργαζομένων ε, διαμεθοριακούς, διαμεθοριακούς με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμεθοριακούς με την Ελβετία. Εκεί λοιπόν το εξή ερώτημα. Οι κανόνες αυτοί θα εφαρμόζονται απευθείας και στην Ελβετία ή θα πρέπει να προηγηθεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία. Κάτι άλλο που μου έχουν αναφέρει ως ανησυχία διάφοροι διαμεθοριακοί εργαζόμενοι είναι το εξή ότι πράγματι η κατάσταση διαφέρει από κράτος σε κράτος. Οι εργαζόμενοι αυτοί σήμερα έχουν κάποια δικαιώματα. Τι θα συμβεί κατά τη μεταβατική περίοδο. Διότι σε τελική ανάλυση η χώρα που θα τους ε, παρέχει ε, τα δικαιώματα, τις παροχές μπορεί να το πράττει υπό συνθήκες λιγότερο ευνοϊκές ε, από αυτές τις οποίες έχουν σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μόνα Σαρτιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τους ομιλητές, ε, τον εισηγητή, τους συνεισηγητές ε, για τα όσα μας είπαν. Αυτή τη στιγμή αναθεωρούμε την οδηγία του 96 για τους απεσπασμένους εργαζομένους και βλέπουμε από, την παρουσίαση που, από τις παρουσιάσεις που είδαμε και από το θέμα των απεσπασμένων εργαζομένων και κυρίως ε, για τις περιπτώσεις εργασίας μικρής διάρκειας ή και της τηλεργασίας όπως αναφέρθηκε ε, όπως βλέπουμε λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν συντονισμό μεταξύ διαφόρων ε, εργασιών δικών μας. Εγώ ανησυχώ. Θα ήθελα να μην υπάρξει ως αποτέλεσμα υπερβολικός διοικητικός φόρτος ούτε απώλεια δικαιωμάτων για τους εργαζομένους. Δεν πρέπει να χαθεί τίποτα. Κατά αυτή την ε, τελική αναθεώρηση αυτόν τον απολογισμό τελικά που θα γίνει τροχρονισμένα. Χρειαζόμαστε και κάποια εργαλεία καταπολέμησης της απάτης φυσικά ε, κυρίως της απάτης των επιχειρήσεων τύπου γραμματοκιβώτια. Ε, η διοίκηση λοιπόν θα πρέπει να προστατεύσει πάνω απ' όλα τους εργαζομένους. Αυτό μας φέρνει όλους εδώ σήμερα και σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι και εγώ είμαι στη διάθεση του εισηγητή ώστε να συντονίσουμε τις εργασίες μας ε, μεταξύ της αναθεώρησης της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους αφενός που πρέπει να συνεχίσει με τη δική της ε, ταχύτητα, με το δικό της ρυθμό ε, αυτό δεν χωρά αμφισβήτηση αλλά που θα πρέπει να συντονίζεται με τις εργασίες του κυρίου Γκίον Παλάς Ευχαριστούμε. Είναι σαφές ότι συνδέονται αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα. Σοφία Λιμπέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία. Και ήθελα να υπογράψω, να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντική η αναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. και είναι πολύ σημαντικό και για τους νέους ε, που πιο εύκολα πέφτουν ε, θύματα αβέβης εργασίας. Δεν πρέπει να μιλάμε λοιπόν μόνο για το παρόν αυτών των νέων αλλά και για το μέλλον τους. Ε, κάποια πράγματα εγώ ομολογώ δεν τα βλέπω πολύ καθαρά. Χρειάζεται, χρειάζεται κάποιες διευκρινήσεις. Εμείς και εγώ φυσικά υπερασπιζόμαστε μια καλύτερη εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων για τον συνυπολογισμό των εισφορών, τον υπολογισμό ε, των κοινωνικών παροχών, των διαφόρων επιδομάτων ε, που λαμβάνουν οι διάφοροι εργαζόμενοι. Αλλά αναρωτιέμαι, σε ποιο βαθμό εδώ θέτουμε υποφυσβήτηση την επικουρικότητα, δηλαδή τις αρμοδιότητες που ανήκουν καθαρά στα κράτη-μέλη. Με άλλα λόγια, τι θα κάνουμε σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ε, θέλει να παρεμποδίσει αυτή την απόπειρα εναρμόνισης που μπορεί να θέσει κίνδυνο για το μέλλον αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέργιο Γκουτιέρες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ και όλους τους ε, ομιλητές σε αυτή την ακρόαση για την ποιότητα των παρεμβάσεών τους. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συνένεση γιατί υπάρχουν διάφορες τάσεις, εντάσεις μεταξύ κρατών μελών. Διότι Πρόκειται για καταστάσεις που βεβαίως ε, αφορούν όλα τα κράτη-μέλη και υπάρχουν ορισμένες κυβερνήσεις που βλέπουν εδώ δυνατότητες πολιτικής αξιοποίησης, ε, εκλογικής αξιοποίησης. Κάποια κράτη-μέλη, λόγω της κρίσης, περιορίζουν τα δικαιώματα ακόμη και των δικών τους των ε, πολιτών όταν ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Η χώρα για παράδειγμα, σε σχέση με την κάρτα περίθαλψης. Και άλλα κράτη-μέλη περιορίζουν την πρόσβαση στις ε, κοινωνικές παροχές για πολίτες άλλων κρατών μελών. Ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Για λόγους ψηφοθυρίας. Είναι λοιπόν ε, αναγκαίο να βελτιωθεί η νομοθεσία για να αποφύγουμε αυτές τις δύο παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών και παραβιάσεις του δικαιώματός τους ε, στην ελεύθερη κυκλοφορία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποια είναι η πολιτική αρχή που είναι η βάση αυτή τη μεταρρύθμισης. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα ή να ε, δώσουμε δίκαιο σε αυτού που τα δημιουργούν. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Βεβαίω χρειάζεται εναρμόνιση. Αλλά υπάρχουν δύο τρόποι εναρμόνιση. προ τα πάνω ή προ τα κάτω. Να λύσουμε τα προβλήματα λόγω ακριβώς ορισμένων ενεργειών ορισμένων που επωφελούνται από τι οικονομικέ και κοινωνικέ συνθήκε. Αυτό είναι το βασικό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιο κράτο πληρώνει. Με ενδιαφέρει να καταλάβω σαφώ τι δικαιώματα χορηγούμε. Δηλαδή, πώ υπολογίζονται οι μήνε που χρειάζονται που για να έχει κανείς δικαίωμα και πώς υπολογίζεται το ύψος των ε, επιδομάτων ποιος είναι ο μέγιστος χρόνος που πρέπει να έχουν εργαστεί και συνεισφέρει πριν έχουν δικαίωμα. Για παράδειγμα, ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι μπορούν να παρέχουν δικαίωμα ε, επίδομα ανεργία για 18 μήνες, άλλα για 6. Το βασικό όμως για το Συμβούλιο είναι ποιος πληρώνει. Εμείς ως Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει τώρα να αρχίσουμε να κάνουμε μικροϋπολογισμούς. Πρέπει να δούμε τι δικαιώματα θέλουμε να αναγνωρίζουμε για τους εργαζομένους δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να μπούμε στον τρόπο σκέψης ορισμένων ε, κομμάτων, σε ορισμένα που όλα αυτά τα χρόνια έχουν περιορίσει τα δικαιώματα των πολιτών τους και άλλων για ακριβώς να κάνουν ψηφοθυρία. Εμένα αυτό που πρόσεξα πολύ είναι ότι αφού ασχοληθήκαμε με τα επιδόματα ανεργίας και βλέπω ότι αυτές, αυτές οι καταχρήσεις αφορούν 27.000 εργαζόμενους σε 500 εκατομμύρια πολιτών της Ένωσης. Πρόεδρος. Και τώρα να ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας για να τους παρακαλέσω καθένα σε 10 λεπτά να απαντήσει. Βλέπετε ότι τα ερωτήματα είναι ορισμένα μεν πιο γενικά για το ποια είναι η γενική σας ε, προσέγγιση της πρότασης της Κομισιόν αλλά και πολύ πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, για λεπτομέρειες. Το βασικό λοιπόν είναι να απαντήσετε σε όλα αυτά γιατί η πρόθεσή μας στη συζήτησή μας αυτή είναι να μας δώσετε την αναγκαία τεκμηρίωση και βοήθεια για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σωστές παρατηρήσεις, σωστές προτάσεις, όσο πιο σωστές γίνεται. Ε, να σας δώσω λοιπόν το λόγο κύριε Άχινχόφερ. Αγαπητέ κυρίε, αγαπητοί κύριοι, με τον συντονισμό των συστημάτων ασφάλισης ε, αρχίζουν όλα. Η πρώτη πράξη του, των κανονισμών 3 και 4 από το 1958 αφορά ακριβώς τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ο, συντονιστός, ο συντονισμός αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο θέμα αυτό ήδη απασχολούσε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1958. Και παρατηρήσαμε ότι οι εξελίξεις ήταν συνεχείς και πάντα υπήρχαν αντιδράσεις αυτές τις εξελίξεις. Πάντα υπήρχαν στοιχεία που προστίθεντο, ε, πάντα υπήρχαν νέα θέματα που προέκυπταν σε διεθνές επίπεδο που ε, απαιτούσαν τροποποίηση και επικαιροποίηση του κανονισμού. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη εξυγχρονισμού αυτού του κανονισμού που άλλαξε τόσο πολύ. Έπειτα, ποιε είναι οι κύριε ιδέε. Οι κύριε ιδέε είναι καταρχά ότι πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία η ελεύθερη μετακίνηση. Πρέπει οι πολίτε να απολαμβάνουν το δικαίωμα τη ε, ελεύθερη μετακίνηση και το δικαίωμα αυτό να ε, προστατεύεται. Και Γι' αυτό θεωρώ πως είναι πολύ καλές οι προτάσεις για την προστασία των ανέργων, για τα επιδόματα ανεργίας. Τώρα, οι αρχές του συντονισμού θεωρώ πως πρέπει ε, να ε, τροποποιηθούν, πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός και ο, η ασφάλιση των ανέργων πρέπει να ε, αλλάξει καθεστώς, να μην ανήκει πια σε αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς. Αυτή η πρόταση είναι σωστή. Τώρα, ο συντονισμός λαμβάνει και μία νέα διάσταση. Η νέα διάσταση έχει να κάνει με την ε, αλλαγή, με την εξαίρεση ορισμένων ε, ομάδων ανέργων. Αυτό θα μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα στο μέλλον. Και υπάρχει αυτό το πισωγύρισμα, όπως είπατε, αυτό όμως που θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ε, πολύ σημαντικό. Χρειάζεται να κοιτάξουμε τις περιπτώσεις ε, που αφορούν διάφορες ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν άτομα τα οποία δεν λαμβάνουν και στην ίδια μου τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια κοινωνικές παροχές ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι, ε, αυτές οι διατάξεις. Υπάρχουν κάποια παραθυράκια που επιτρέπουν στην νομοθεσία να το κάνει. Τώρα, η νομοθεσία για τους ανέργους πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Πρέπει να γίνουν ε, έντονες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να αφορούν πρώτον την ενίσχυση της ελεύθερης μετακήρυσης και δεύτερον ε, τα δικαιώματα των μετακινούμενων εργαζομένων. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν και το θέμα της εξαγωγής των ε, επιδομάτων των κοινωνικών παροχών, να δούμε υπό ποιε ε, συνθήκες αυτό γίνεται. Σε γενικές γραμμές θεωρώ καλό να υπάρχει αυτή η προστασία. Τώρα, εδώ και πάρα, πολλές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε δει ότι το κράτος το οποίο φιλοξενεί εκείνη την στιγμή όποιον αναζητά εργασία είναι υπεύθυνο και για την καταβολή των ε, επιδομάτων ανεργίας και διάφορων άλλων ε, κοινωνικών παροχών. Ε, δεν είναι χρήματα κάποιου άλλου κράτους, είναι χρήματα του κράτους το οποίο διαμένει εκείνη τη στιγμή ο εργαζόμενος. Ε, η ελεύθερη μετακίνηση είναι σημαντική βέβαια για εκείνους που ήδη έχουν κάποια εργασία, ακόμα σημαντικότερη όμως για εκείνους που την αναζητούν γιατί διευρύνονται έτσι οι δυνατότητες απασχόλησής τους. Και φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις οικογενειών ή συντρόφων όσων ε, αλλάζουν χώρα για να εργαστούν, οι οποίοι ακολουθούν και πρέπει να βρουν και εκείνη κάποια μορφή απασχόλησης. Τώρα, η περίπτωση της Ελβετίας. Ε, πράγματι, η Ελβετία πρέπει να συμπεριληφθεί, αν όχι άμεσα σύντομα τουλάχιστον, στο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και φυσικά πρέπει να, γίνει, να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ε, πρόοδου και της εφαρμογής. Τώρα, η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων δεν ε, συμπεριλαμβάνεται στην ε, αναδιατύπωση της πρότασης. Και αυτό γιατί δεν ανήκει άμεσα σε θέματα συντονισμού ε, να αφαιρθώ επίσης στο άρθρο 5 του ε, κανονισμού, όπου αναφέρεται στα παιδιά. Τα παιδιά ε, τα οποία ζουν σε άλλος, άλλο κράτος μέλους από εκείνο το οποίο καταβάλει τις ε, διάφορες παροχές και τα οποία εξαιρούνται από αυτές. Εδώ πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης έτσι ώστε να αποφευθούν οι διακρίσεις, να μην ανήκουν λοιπόν τα παιδιά σε κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς. Χρειάζεται και εδώ καλύτερος έλεγχος και σίγουρα ε, προσπάθεια για να μην αυξηθεί υπερβολικά η γραφειοκρατία. Όμως, όπως σας είπα, ε, αυτό δεν ανήκει στο νηφιστάμενο κανονισμό, στο, στην αναδιατύπωση. Βλέπω τώρα πράγματι κάποια πλεονεκτήματα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα για τις προθεσμίες και τα ανώτατα ε, διαστήματα. Θεωρώ πως είναι λοιπόν καλή η πρόταση εκεί, διότι υπάρχει προσπάθεια να γίνει μια προσέγγιση προσέγγιση της ε, νομοθεσίας των διάφορων ε, κρατών μελών έτσι ώστε να υπάρχει και μια εξίσωση των ε, κοινωνικών παροχών, επιδόματα ασθένειας για παράδειγμα, ανεργίας κτλ. Σίγουρα βέβαια δεν πρέπει να υπερβούμε των αρμοδιοτήτων μας. Τώρα, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα παράτασης πέρα από το χρονικό όριο των ε, δύο ετών. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται να εξεταστούν οι διάφορες δυνατότητες που ε, απορρέουν από το άρθρο 16 που αφορά τη, τους ανέργους. Τώρα, ε, για τους διαμεθοριακούς εργαζόμενους, θα επαναλάβω ότι το πρόβλημα με τους διαμεθοριακούς εργαζόμενους είναι το εξής. Σύμφωνα με το υφιστάμενο δίκαιο, όταν κάποιος μένει άνεργος, πρέπει να, μετα... την χάνει μεταχείριση ανέργου που έχει μείνει άνεργος στο ε, κράτος που διαμένει, όχι στο κράτος που εργάστηκε. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει εργαστεί σε ένα άλλο κράτος, πρέπει να θεωρείται ότι έχει μείνει άνεργο σωστό κράτος που μένει. Χρειάζεται βέβαια εδώ να αποδειχθεί αυτό. Τώρα αναφέρθηκε επίσης και το θέμα της επικουρικότητας. Νομίζω πως εδώ δεν τίθεται θέμα επικουρικότητας. Η επικουρικότητα έχει να κάνει με την κατάρτιση του συστήματος, ε, με, ε, τη, με τον καθορισμό του ύψους των ε, παροχών, των συντάξεων κτλ η εθνική νομοθεσία έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και η επικουρικότητα εδώ δεν πρέπει να συγχαίει τα πράγματα. Τώρα, ε, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο συντονισμός είναι απαραίτητος και είναι μάλιστα πιο χρήσιμος ή καλύτερος από οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε εθνική νομοθεσία. Τώρα, ε, για τους μη ε, ενεργούς οικονομικά που έχουν ανάγκη, χρειάζεται ε, μεγάλη προσπάθεια, διότι με την αυτόνομη ρύθμιση κάθε κράτους μέλους για αυτήν την ομάδα ανθρώπων κινδυνεύουν να μείνουν εκτός κοινωνικού συστήματος, εκτός κοινωνικής προστασίας αυτοί οι άνθρωποι διότι υπάρχει ο κίνδυνος όποιος ε, δεν έχει κοινωνικές, ε, κοινωνική προστασία σε ένα κράτος να μεταβεί σε άλλο και να μην έχει ούτε εκεί. Η πρόταση λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό και ε, δείχνει ότι η έλλειψη συντονισμού, ευρωπαϊκού συντονισμού οδηγεί, θα οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα, σε αποκλεισμό ομάδων ανθρώπων όμως ε, είναι κάτι που παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρέπει ε, να συμπεριλάβει την ομολογία. Δεν υπάρχει όμως μεγάλη σαφήνεια σε αυτόν τον τομέα, το πώς θα γίνει αυτό. Και για το συντονισμό να αναφέρω και κάτι στο τέλος, ότι θα ότι με την ε, ελεύθερη μετακίνηση επικεντρωνόμαστε μόνο σε όσους ε, αναζητούν εργασία σε όσους ήδη εργάζονται και αλλάζουν χώρα και όχι σε αυτούς που, ονομάζουμε, σε αυτούς που κάνουν αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό τουρισμό, στους μη ενεργούς οικονομικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο και ελπίζω να αντιμετωπιστεί με το σωστό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Ντεγιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις, ε, ε, πολλές ε, και διαφορετικές, διαφορετικής φύσης. Ξεκινώντας από μια ερώτηση που ακούσαμε ότι καθώς κοιτάμε το σύνολο της πρότασης της Κομισιόν αν είναι καλή. Διότι φυσικά στις προτάσεις που κάναμε φάνηκε να κρατάμε κάποια απόσταση από το κείμενο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι αλλαγέ αλλαγές ε, ουσιαστικά είναι καλές ως προτάσεις. Όπως είπα και νωρίτερα και είπαν νωρίτερα και συναδελφοί μου, ε, κοιτώντας τα βασικά στοιχεία πρέπει κανείς ε, να το ψάξει λίγο περισσότερο, να δει τις λεπτομέρειες και να αναζητήσει, να δει ποιες θα είναι οι συνέπειες εντό του πολύ, μέσα από αυτό το πολύ τεχνικό κείμενο, ε, συμφωνώ μαζί σα. Ποιε θα είναι λοιπόν οι καθημερινέ συνέπειε, ε, οι συνέπειε στην καθημερινότητα του κόσμου. Εκεί ε, θα μπορέσουμε να βρούμε κενά και να θέσουμε ερωτήματα για το κατά πόσο το προτείνομενο κείμενο πράγματι θα φέρει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Ε, όσον αφορά τις παροχές ανεργίας, τα επιδόματα ανεργίας, ε, στα οποία αφιέρωσαμε και τον περισσότερο χρόνο για τους διαμεθοριακούς ε, εργαζομένους, η αλλαγή αυτή, όπου το τελευταίο κράτος απασχόλησης θα έχει την αρμοδιότητα καταβολής των επιδομάτων ανεργίας, είναι, όπως είπα, λογικό βήμα. Όπως κάποιο από σας είπε, μάλιστα, το κράτος αυτό στο οποίο έχουν καταβληθεί οι κοινωνικές ε, εισφορές, ε, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Ε. Είναι πολύ λογικό να καταβάλει και τα επιδόματα ενεργείας. Ωστόσο πιστεύω ότι πρέπει να δει κανεί στο κείμενο αυτό προτείνεται με αυτή την εισαγωγή διαφορών περιόδων 12 μηνών, περισσότερο, λιγότερο, τριών μηνών και να αναρωτηθεί λοιπόν μήπως το κείμενο αυτό το οποίο ήδη είναι δύσκολο ε, στην κατανόηση όπως και το σημερινό βέβαια μήπως τελικά μήπως απλά δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση για ένα δημοσιογραφικό εργαζόμενο, ο δεν θα καταλαβαίνει ποια είναι τα δικαιώματά του. Ε, οπότε ίσως ε, εγώ θα πρότεινα να βρίσκαμε έναν ε, πιο απλό τρόπο διατύπωσης που να δίνει απαντήσεις στις διάφορες ερωτήσεις. Έχουμε αυτή την περίοδο των 12 μηνών, είναι διαδοχική, σπαστή, πώς, πώς γίνεται. Κάποιο μέλος είπε πώς θα υπολογίσουμε τους τρεις μήνες, όταν κάποιος ξεκινάει ας πούμε την καριέρα του μπορεί να εργάζεται περιστασιακά αρχικά και πώς έτσι λοιπόν θα αποκτήσει το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας. Για να προέσω τώρα σε μια άλλη ερώτηση. Ο κανονισμός για την κοινωνική ασφάλιση ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός πρόωθησης της ελεύθερης ε, κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτή την έννοια, αυτό που ανέφερα και νωρίτερα και για το οποίο ακούσαμε μια ερώτηση, οι διοικητικές διατυπώσεις που απαιτούνται ώστε ε, διασφαλίζουν ότι κάποιο ε, που σύμφωνα με τον κανονισμό υπόκειται σε ένα συγκεκριμένο σύστημα κοινωνική ασφάλιση πράγματι καταβάλει τι ε, συνεισφορέ αυτέ. Και δεδομένου ότι πρέπει να προωθήσουμε αυτή την ελεύθερη κυκλοφορία, κατά πόσο λοιπόν σε αυτέ οι διοικητικέ διατυπώσει θα προστεθούν. Διότι αλλιώ ε, στο διεθνές περιβάλλον που βρισκόμαστε σήμερα οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν να επιτρέπουν στον κόσμο να εργάζεται διεθνώς. Εάν έχουν μια, ένα απλό καθεστώς ε, διαμεθοριακού εργαζομένου, ε, εάν κάποιος μένει στο κράτος Α και εργάζεται στο Β και εργάζεται ας πούμε με μερική απασχόληση, αυτό είναι συνήθες στις κάτω χώρες. Αν εργάζομαι σπίτι μου λοιπόν τη μία ημέρα τη βδομάδα μόνο, μιλάμε για το 25% ε, αλλαγή δηλαδή στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη δική μου χώρα, σε αυτή την περίπτωση, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις ε, τις οποίες πρέπει να υποστεί η επιχείρηση, κάτι που δυσχεραίνει ουσιαστικά την απασχόληση κάποιου εργαζομένου. Αυτό που φοβάμαι λοιπόν ότι ε, θα εμφανιστεί κάποια τάση απαγόρευσης να εργάζεται κάποιο ε, στο σπίτι με τηλεργασία. Ενώ δεν είναι αυτό ο σκοπό του κανονισμού. Ο σκοπό του κανονισμού είναι ο κόσμο να μπορεί να επιτρέπεται να εργαστεί ε, σε πολλές χώρες. Και φυσικά το νομικό κείμενο το επιτρέπει, αλλά η πρακτική εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο με διάφορους τρόπους. Μια άλλη ερώτηση που ακούσαμε για την τηλεργασία. Πράγματι η τηλεργασία θα αποτελεί όλο και συχνότερο φαινόμενο στο μέλλον. Ε, ειδικότερα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας. και των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίε πρέπει να εξελιχθούν ώστε να συνεχίσουν αυτές οι μορφές απασχόλησης ε, από τους εργοδότες, γιατί ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις ε, που ξέρω εγώ, ας πούμε, θέλουν να συμμορφώνονται με του κανονισμού κοινωνική ασφάλιση, να ασφαλίζουν τους ανθρώπους σωστά, στη σωστή χώρα και αυτό συμφέρει και τους εργαζομένους ε, γιατί είναι άσχημε οι συνέπειε σε περίπτωση που κάποιος είναι ασφαλισμένος στη λάθος σύστημα κοινωνική ασφάλισης και πάθει κάποιο ατύχημα και χρειάζεται ιατρική περίθαλψη. Ε, σε περίπτωση που έχει ασφαλιστεί σε λάθος χώρα θα πρέπει λοιπόν να διευκολυνθεί αυτή η κατάσταση. Και αυτό θα βοηθήσει και στην καταπολέμηση τη απάτη. Διότι εφόσον υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός, ο οποίος διασφαλίζει ότι οι κοινωνικές φορές πληρώνονται, καταβάλλονται στις σωστές αρχές, ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να εξετάσει και κατά πόσο έχει καταβληθεί το σωστό ποσό. Πολλές ερωτήσεις δηλαδή που ακούσαμε σήμερα και πολλές λεπτομέρειες ε, που ακούστηκαν ε, θα πρέπει να εξεταστούν ε, κατά την πιο τεχνική εξέταση του κειμένου κατά άρθρο που να δούμε, ε, θα δούμε τι ζητήματα προκύπτουν από το πρωτονομικό κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κάρλος Καρθία. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, όταν εξετάζω τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα ε, μου έρχονται δύο ή μάλλον δυόμιση επιτεύγματα. Πρώτον, το έρασμος. Δύο, η Ευρωπαϊκή ε, Κάρτα Περίθαλψης. Το μισό επίτευγμα ε, είναι το ευρώ. Τώρα ίσως θα έλεγα ότι είναι ένα τέταρτο. Αλλά αυτά είναι τα μεγάλα επιτεύγματα που καταλαβαίνει ο πολίτης. Με ρώτησε η ευρωπαικη καρτα περιθαλψης το μισο επιτευγμα ειναι το ευρω τωρα πώς εκτιμώ την πρόταση στο σύνολό της. Θα είμαι σαφής. Εμένα μου αρέσουν οι κανονισμοί συντονισμού και γι' αυτό υποβάλλω επικρίσεις. Γιατί θέλω να είναι άψογοι οι κανονισμοί. Αν με ρωτήσετε σε τι ποσοστό συμφωνώ με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έλεγα 80%. Εντάξει. Οι επικρίσει μου είναι επικοδομητικέ. Θα ήθελα να είναι τέλεια. Ε, είμαι ερωτευμένο με αυτού του κανονισμού και θα ήθελα λοιπόν να είναι όμορφοι και τέλειοι. Ε, αν ε, ε, μου πει ε, τι πρέπει ε, να κάνουμε αν ε, η επιλογή είναι μεταξύ απόρριψης και έγκρισης. Θα έλεγα, ε, με επιφυλάξεις ε, τον εγκρίνω. Τώρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση μου έγινε. Τι δυνατότητες και τι βελτιώσεις έχουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε, ούτως ώστε να υπάρχει εξαγωγή του επιδόματος ενεργείας μέχρι 6 μήνες. Ίσως να σε εκπλήξει η απάντησή μου. Πριν από λίγο, στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του Δεκεμβρίου, η Ισπανή, Ισπανίδα υπουργό είπε το εξή. Αυτές οι παροχές όταν τις ε, εξάγουμε για λιγότερο από τρεις μήνες καταφέρνει να ενταχθεί ο εργαζόμενος στην άλλη χώρα σε ποσοστό λιγότερο από 10%. Εάν κάνουμε αυτές τις παροχές για 6 μήνες, η πιθανότητα ένταξης των εργαζομένων είναι 70%. Η Ισπανία είναι η τρίτη χώρα από πλευράς αριθμού εργαζομένων που είναι σε άλλες χώρες. Δηλαδή, μάλλον αντίστροφα. Έχουμε ε, πολλές, πάρα πολλού εργαζόμενους από τι άλλε χώρες της Ένωση. Στην ε, Ισπανία έχουμε μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων από άλλες χώρες. Άρα αυτή η εξαγωγή δεν βοηθάει μόνο το άτομο αυτό προσωρινά, το βοηθάει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας της χώρας όπου εργάζεται. Τρίτον, κοιτάξτε, καταλαβαίνω απόλυτα τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αναφέρθηκα στην απόφαση για το Ηνωμένο Βασίλειο που ε, δημοσιεύθηκε 7 μέρες πριν από τον Brexit. Είναι μια πολιτική απόφαση. Δεν ξέρω εάν ε, έπρεπε να εκδοθεί τώρα η απόφαση, ε, θα εκδίδεται το ίδια. Πρέπει λοιπόν να την εξετάσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλύτερα θα ήταν να την αγνοήσουμε σε μεγάλο βαθμό. Όλες οι υπόλοιπες, όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις δεν αναφέρονται σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Στρίκτο σένσου. Τις αποκαλούν οι ειδικέ μικτές παροχές όπου δεν εισφέρει ο εργαζόμενος. Θα μου πείτε, μα είναι το ίδιο. Ή ε, απλώς συγκρίνουμε την ε, κοινωνική πρόνοια με την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ε, παροχές που δίδονται σε αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη. Είναι επίσης ε, ε, περιπτώσεις όπου δίδεται απλώς κάποιο συμπλήρωμα. Δεν είναι οικογενειακό επίδομα, δεν είναι σύνταξη. Είναι συμπληρωματικές παροχές πολύ ειδικέ. Να είναι σαφές αυτό. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνει παραπέρα από αυτά τα οποία έχει ορίσει το δικαστήριο και θα μπορούσε να είναι ένα ε, ιδιαίτερα αποτελεσματικό όργανο για να προωθήσει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Εγώ δεν είμαι υπέρ της ε, κατάχρησης και των ε, απατών. Φυσικά πρέπει να τα καταπολεμήσουμε. Αλλά όπως λέμε στην Ισπανία, δεν είναι δυνατόν να σκοτώσουμε κουνούπια με κανονιές. Μου μιλήσατε για την απασχόληση και την ανεργία μάλλον. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσουμε στο εξή πιστεύω. Εάν εγώ συνάψω ε, μία σύμβαση μαζί σας, τότε πρέπει να ε, με πληρώσετε. Για να μπορέσω και εγώ να πληρώσω τους άλλους με τους οποίους έχω συμβάσεις. Εάν πληρώνω λοιπόν φορές, τότε και εσείς πρέπει να μου δώσετε τις παροχές, το επίδομα ανεργίας. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω είναι να πληρώσω εγώ κάποιον και μετά να με πληρώσει κάποιο τρίτο το επίδομα ανεργία. Μόνο και μόνο επειδή διαμένω σε κάποια χώρα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ενιαία λύση. Πρέπει να βρούμε ένα στοιχείο συντονισμού. Γιατί κοιτάξτε, αν πω εγώ στο φουρναρί μου, κοίταξε, εσύ εργάζεσαι στη Γερμανία, αλλά θα σε πληρώσει η Ισπανία, δεν θα το καταλάβει. Και αυτό που είναι σημαντικό, που πρέπει λοιπόν να περιέχει ο κανονισμό, είναι να είναι κατανοητό. Και αυτό είναι, αυτός ο κανονισμός είναι δυσνόητος. Τώρα για το θέμα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Τώρα αυτό θα είναι πραγματικά σαν, την, σαν να ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Κοιτάξτε, και πού θα πρέπει να λάβει τα επιδόματα, για παράδειγμα, να λάβουν τα επιδόματα τα παιδιά ενός συνταξιούχου. Πού? Στην Ισπανία που μένει ο συνταξιούχος ή στη Γερμανία που μένουν τα παιδιά. Πώ ακριβώ θα το πληρώσουμε. Στην ουσία καταργούμε τη δυνατότητα συντονισμού, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Α ε, σκεφτείτε πώ είναι η κατάσταση σε μια χώρα στην Ισπανία, που πληρώνουμε πολύ μικρά επιδόματα για τα παιδιά. Αν τα παιδιά μας μείνουν στη Γαλλία, αν πρέπει να πληρώσουμε τα γαλλικά οικογενειακά επιδόματα, τότε θα καταρρεύσει το σύστημα κοινωνική ασφάλισης. Πώ θα πληρώσουμε σε κάποια άτομα που ζουν ε, εκτός Ισπανίας περισσότερα από όσους πολίτε μα ζουν εντό τη Ισπανίας. Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι απλοί οι κανόνε και να είναι κατανοητοί. Τώρα, αναφερθήκατε στην Ελβετία. Αν εγκριθεί αυτός ο κανονισμός, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε. Στην Μικτή Επιτροπή Ευρώπης Ελβετίας και αν συμφωνήσει η Ελβετία θα πρέπει να το εφαρμόσει και για του διαμεθοριακού εργαζόμενους στην περίπτωσή τη. Κάλυψη ασφάλισης, ε, συγγνώμη, κάλυψη ε, ασθενείας. Να σα εξηγήσω το εξή. Το δικαστήριο αντιμετώπισε μια υπόθεση ασφάλισης εξαρτωμένων μελών και είπε πού ακριβώς θα μπει στον κανονισμό και είπε επειδή δεν αναφέρεται επειδή δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στον κανονισμό, δεν αναφέρεται η ασφάλιση εξαρτωμένων πουθενά, το βάλαμε στην ασφάλιση ασθενείας. Αλλά δεν υπήρξε αμοφωνία γι' αυτό στο Συμβούλιο, έγιναν διαπραγματεύσει, τρία κράτη διαφωνούσαν και τελικά συμφώνησαν και συμπεριλήφθηκε στην ασφάλιση ασθενεία το θέμα των επιδομάτων για τα εξαρτώμενα μέλη. Τώρα ένα από αυτά τα τρία μέλη θα φύγει από την Ένωση, από τα κράτη-μέλη που διαφωνούσαν, οπότε υπάρχει ειδική πλειοψηφία. Βέβαια, πιο λογικό θα ήταν να δημιουργηθεί χωριστή τέτοια κάλυψη, σε ένα χωριστό κεφάλαιο, όπου θα διτηρηθούν βέβαια οι προηγούμενες διατάξεις, κατά 90%. Νομίζω πως είναι θέμα καθαρά ε, τεχνικό ε, νομικό. Νομικό λοιπόν. Τώρα, πώς θα συνδεθεί αυτός ο κανονισμός με την οδηγία για τους αποσπασμένους. Κοιτάξτε, ε, πολύ καλύτερα έχουν αποτελέσματα οι κανονισμοί από τι οδηγίες. Τώρα έχουμε μια πρόταση οδηγία που θα τροποποιήσει την προηγούμενη. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και να δούμε αν μέσω αυτής της νέα οδηγίας θα έχουμε δυνατότητα κάπως να την ε, συνδέσουμε με τον κανονισμό. Αλλά το βασικό είναι να συνεχίσουμε όπω κάναμε και στο παρελθόν. Και με επιτυχία. Τώρα, για να τελειώνω εφαρμοστικέ και εκτελεστικές και κατοξιοδότηση πράξη. Αλλά υπήρξε μία έκθεση της Γαλλικής Γερουσίας που είπε ότι οι εκτελεστικές παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητα. Γιατί οι εκτελεστικές πράξεις που εφαρμόζει η Κομισιόν δεν ελέγχονται από τεχνικά κοινοβούλια. Αλλά υπάρχει και κάτι παραπάνω. Αυτή είναι μια διαμάχη στην οποία δεν θέλω να εισέλθω. Είναι θεσμική διαμάχη που έχει πολύ ευρύτερε διαστάσει. Η γενικότερη αντιμετώπιση αυτών των δύο ειδών πράξεων. Αλλά να σα δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάρετε την πρόταση αυτή κανονισμού, λέει δίδεται η αρμοδιότητα στην Κομισιόν να διατυπώσει και να εγκρίνει τα παραρτήματα του κανονισμού. Δηλαδή, αν διαβάσετε αυτά τα παραρτήματα, θα έχετε μεγάλα προβλήματα, είναι ιδιαίτερα δυσνόητα. Αλλά υπάρχει ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα συγγνώμη, το παράδειγμα 3, όπου λέει το οποίο λέει κάτι το οποίο ευτυχώς το Κοινοβούλιο υποχρέωσε το Συμβούλιο να δεχθεί. Γιατί έτσι έχουμε κάποια δικαιώματα για τους εργαζομένους και για τους πολίτες και για τα παιδιά των μεταναστών εργαζομένων. Δηλαδή καταφέρατε να έχουν κάποια δικαιώματα μόνιμα. Με αυτές τις εκτελεστικές και καταξοδότηση πράξη θα χάσετε όμως μια σειρά από δυνατότητες και αρμοδιότητες. Γιατί τα παραρτήματα ή τουλάχιστον ορισμένα έχουν ε, τόση αξία όσο και το κείμενο του κανονισμού. Όταν εφαρμόζουμε τον κανονισμό, τον εφαρμόζουμε με βάση και τα παραρτήματα. Άρα, Εάν δώσετε στην Κομισιόν την αρμοδιότητα για όλα αυτά τα θέματα, θα γίνονται πολύ σύντομα τα πράγματα, αλλά θα έχετε χάσει πολλέ δυνατότητε ελέγχου. Θα μου πείτε, ναι, εντάξει, μπορούμε να το απορρίψουμε. Αλλά όχι, εγώ δεν θέλω να απορρίψετε, ε, θέλω να διαπραγματευτείτε. Όπω κάνατε και με τον κανονισμό του 2010 και για την αρχή τη επικουρικότητα. Νομίζω ότι στο 99% των περιπτώσεων ο μηχανισμός αυτός ε, βεβαίως ε, έχει έννοια αλλά τα θέματα που τίθενται στη Γαλλία είναι πολύ περίπλοκα, πολύ ε, ενδιαφέροντα, αλλά πολύ περιορισμένα. Ανησυχούν πολύ για την οδηγία της απόσπασης και άρα κάθε στιγμή, για κάθε θέμα πρέπει να αναφέρονται και σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κύριο Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους τρεις εμπειρογνώμονες οι οποίοι πιστεύω μας έκαναν ε, μια ε, διεξοδική ανάλυση της πρότασης. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ σε αυτά που ακούσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι αν άκουσα καλά και οι τρεις εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η πρότασή μας είναι καλή. δεν λέω ότι δεν πρέπει να την αλλάξουμε, αλλά ε, ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ε, όπως φαίνεται μας λένε ότι συμπεραίνουν πως ε, έτσι έχουν τα πράγματα. Φυσικά θα πρέπει να συνεργαστεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, όλοι μεταξύ τους ώστε οι συνομοθέτες να καταλήξουν σε ένα νομοθέτημα ικανοποιητικό. Με δύο λόγια ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των εργαζομένων και του κράτους όπου έχουν εργαστεί. Αυτό σχετίζεται με τα επιδόματα ανεργία. Αυτή είναι μια πτυχή και θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν δημιουργούμε νέα δικαιώματα εδώ. Δεν αναγκάζουμε τα κράτη-μέλη να παρέχουν επιδόματα ενέργεια μετά από τρει μήνε. Λέμε ότι μόνο μετά από τρει μήνε θα μπορεί ένα κράτο μέλο στο οποίο έχει ε, μεταφερθεί ένα ε, εργαζόμενο να δώσει επίδομα ενέργεια. Απλά δεν υποχρεώνουμε κάποιο κράτο ε, να δώσει κάτι περισσότερο σε έναν μετακινούμενο εργαζόμενο σε σχέση με αυτό που βρίσκεται ήδη εκεί. Αυτό είναι το ένα όσον αφορά την αγορά εργασία. Το δεύτερο είναι το ζήτημα των καταχρήσεων. Ε, πράγματι, το ζήτημα αυτό αναφέρθηκε από πολλού, είναι ευαίσθητο ε, και ακαθόδε. Πρέπει κανείς να είναι σίγουρος ότι δεν ε, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης οι ευρωπαϊκοί κανόνες για λόγους απάτης. Αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουμε να έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες που να δυσχεραίνουν την ε, ελευθερία κυκλοφορία. Και εκεί αναφέρομαι και στα ζητήματα τη ίση μεταχείριση των μη ενεργών ε, εργαζομένων. Να σα διαβεβαιώσω ότι οι μη ενεργοί δεν. Ε, σε αυτή την περίπτωση ενεργών δεν συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη της οικογένειας. Δυναμή του κανονισμού Ε, διατηρείται ο, εργαζόμενος, ε, διατηρείται η έννοια του εργαζόμενου ε, και δεν θέλω να μπω και σε μεγάλη ανάλυση με τον Κάρλος, ο οποίος μάλιστα είναι ο μόνος στην Ευρώπη που μπορεί να μιλήσει όμορφα για τον, για τον κανονισμό 883 δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε πιο πέρα από την κωδικοποίηση. έχουμε υπερβάλει με την κωδικοποίηση, εμεί κωδικοποίησαμε τι αποφάσει. Ε, μία απόφαση. Υπάρχουν και άλλε πολλέ αποφάσει. Ε, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε ούτω ή άλλω και στο Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν. Αποφύγουμε τι ε, καταχρήσει και τι απάτε χωρί να θέτουμε εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία. Το τρίτο θέμα είναι οι περιπτώσει απάτη. Ε, η κατάχρηση και απάτη δεν είναι το ίδιο. Ε, στις περιπτώσεις της απάτης, ε, ουσιαστικά τις απάτης έχουμε στον τομέα της απόσπασης εργαζομένων. Θέλουμε λοιπόν να αναγκάσουμε τις εθνικές αρχές ε, να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους ώστε να διασφαλίζουν ότι θα μπορούν να εντοπίσουν τις περιπτώσεις ε, όπου κάποιο ε, δεν έχει ε, εγγραφεί στο σύστημα κοινωνική ασφάλιση μια χώρα, στο να εφαρμόζεται ο νόμος ουσιαστικά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσω τη ενίσχυση τη συνεργασία. Και τέλος έχουμε και το θέμα τη Αφήνεια. Όπω είπατε το δίκαιο μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εφόσον το καταλαβαίνει κανεί. Αυτό είναι και ο σκοπό μα Γι' αυτό θέλουμε να το κεφάλαιο για τις τη μακροχρόνια φροντίδα υγεία. Αυτή για την πρότασή μα Να σα υπενθυμίσω ότι ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορούμε να συζητήσουμε με εσά και με το Συμβουλίο ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το θέμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Τόσο σημαντικό που στην ε, ε, κοινή διακήρυξη Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιών δίνεται προτεραιότητα στο θέμα αυτό όπου εμείς δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε τάχιστα με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας Γκυγιον ε, εισηγητής. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν σημαντικό, γι' αυτό έκανα αυτή την ερώτηση τόσο απότομα. Ε, ήταν σημαντικό, θεωρούσα, να μάθουμε ποια είναι η συνολική, η γενικότερη εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων ε, όσον αφορά την πρόταση αυτή. Και πιστεύω ότι σήμερα καταφέραμε να ορίσουμε κάπως το πλαίσιο της πρότασης αυτής, της πρότασης αναδιατύπωσης του κανονισμού. Όπως βλέπουμε, σήμερα έχουμε μια πρόταση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει ε, τις συνθήκες κυκλοφορίας των εργαζομένων με μεγαλύτερη προστασία των συμφερόντων του. Ταυτόχρονα όμως, ε, παρατηρούμε ότι στην πρόταση αυτή μπορεί να υπάρξουν παρενέργειε για να τι ονομάσουμε έτσι, που να μειώσουν ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα ε, και τι οποίε πρέπει να μειώσουμε. Ε, Θέλω να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στο εξή ζήτημα. Ε, για τι επιχειρήσει, για τη διοίκηση και για του ε, εργαζομένου δεν πρέπει να γίνει υπερβολικό ο διοικητικό φόρτο ούτε να δημιουργεί ανισότητε μεταξύ των δικαιούχων γιατί αυτό τελικά μπορεί να γίνει. Ε, και μετά ουσιαστικά κανεί δεν θέλει να απολαύει αυτών των δικαιωμάτων διότι είναι υπερβολικά περίπλοκο. Αλλά αυτό που θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και θα το κάνουμε με μεγάλη προσοχή, ειλικρίνεια και προσπαθώντας να βρούμε κάποιο συμβασμό μεταξύ μας το θέμα των ανενεργών ε, εργαζομένων. Αντιλήφθηκα πού είναι το προβληματάκι, που, τι θα μπορούσε ουσιαστικά να ανατρέψει το όλο ζήτημα, ε, να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι που θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Γι' αυτό θεωρώ ότι απόψη μεθόδου τώρα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα και στρέφουμε τώρα προς τους όλες καθώς και προς τους συνεισηγητές ε, για το θέμα των αποσπάσμενων εργαζομένων για να προτείνω το εξή. Πρώτον, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα εργασίων το οποίο θα πρέπει να στάλει πριν το καλοκαίρι και να είναι σαφές για το σύνολο της ε, Επιτροπής ε, να γνωρίζουμε από σήμερα το χρονοδιάγραμμα της ημερομηνία και την προοπτική τελική συμφωνία επί του θέματος. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη πρόταση θα είναι να γίνει και μια πρόταση να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε όχι μόνο με εμπειρογνώμονες και ειδικότερα τους τρεις που έχουμε εδώ μπροστά μας, αλλά και με διάφορους άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, να σκεφτούμε τους εκπροσώπους εργαζομένων, επιχειρήσεων, αλλά όχι μόνο, ε, ίσως και άλλους, γιατί όχι εκπροσώπους από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλειας των διαφορών χωρών και η άποψή τους είναι σημαντική. Και με αυτό το σκεπτικό έχω να κάνω μια, θα κάνω και εγώ μια, κάποιες προτάσεις ε, για να γίνουν κάποιες περιορισμένες συναντήσεις με τους συνεισηγητές, με τους σκιώδεις ε, και κάποια ταξίδια εργασίας ώστε να πάμε να επισκεφτούμε ορισμένες χώρες για να καταλάβουμε πολύ καθαρά τις σημαντικές διαφορές θα πάρουμε κάποιες χώρες ε, ε, παραδείγματα μεταξύ εισαγωγικών, κάποιες χώρες ε, αντιπροσωπευτικές αναπεριοχή. Για παράδειγμα μια χώρα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μια χώρα της Βόρειας, μια χώρα της Νότιας Ευρώπης, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και να καταλάβουμε καθαρά ποιες είναι οι δυσκολίες και ειδικότερα ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες Επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει και κάποια ε, μελέτη προκατακτική του μεταναστευτικού ζητήματος, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό το ζήτημα σαν να μην υπάρχει. Σε κάποιες χώρες σήμερα υπάρχει εσωτερική ενδευρωπαϊκή μετανάστευση και άλλες που δέχονται μετανάστες ε, από αλλού. Εάν, ε, όπως σχέση Ισπανίας-Γερμανίας ας πούμε, υπάρχει... Πρέπει να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Αυτά είχαν από σήμερα κύριε Πρόεδρε, οπότε μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει μια πρώτη πρόταση χρονοδιαγράμματος και μεθόδου εργασία που θα σταλεί σε όλους τους και συζητητές της ομάδας και στους συνσηγητές για το θέμα των αποσπασμένων εργαζομένων γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οπότε κλείνουμε αυτή μας την ε, ακρόαση. Νομίζω ότι μέσω των ε, παρεμβάσεων που ακούσαμε είτε των ομιλητών είτε των συναδέλφων καθίσταται σαφές ότι έχει στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης το θέμα αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που είναι στην καρδιά της ουσίας της ελεύθερης κυκλοφορίας, της κινητικότητας είτε της διαμεθοριακής, είτε απλώς από μία χώρα στην άλλη και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η κινητικότητα σε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της καθημερινότητας των ανθρώπων, την ανεργία, την υγεία, τις συντάξεις, ε, τα κοινωνικά επιδόματα, τα οικογενειακά επιδόματα. Τίθενται πολλά ερωτήματα και για τη διατήρηση κάποιων δικαιωμάτων, αλλά και για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι δυνατότητες κατάχρησης και απάτης. Ε, διαπιστώνουμε ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Αλλά περιπλοκότητα δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να επιδιώξουμε τα πιο ευδιάκριτα, τα απλούστερα, τα πιο διαφανή μέτρα. Γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι αναπόφευκτα θα είναι αναποτελεσματικά. Και κάτι άλλο που το υπογράμμισαν πολλοί ομιλητές και στην τελευταία παρέμβαση του εισηγητή μας, η απόλυτα αναγκαία σύνδεση της εργασίας μας για το θέμα αυτό, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, με την εργασία για την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση. Γιατί είναι προφανής οι ε, ομοιότητες μεταξύ αυτών των δύο θεμάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι και ο εισηγητής μας και οι σκιώδεις έχουν επαρκές υλικό για να εργαστούν. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά θερμά πέρα από μια τυπικότητα, όχι, πολύ ουσιοδός. Ευχαριστώ πολύ τους ε, ειδικού μας για την συμβολή τους, για τις αρχικές του παρουσιάσει, αλλά ιδιαίτερα για την υψηλή ποιότητα των απαντήσεών τους στις ερωτήσεις. Και το θέμα αυτό βεβαίω δεν είναι τόσο σεξι, για να το πω έτσι, αλλά μέσω των παρεμβάσεών σας όντω καταφέρατε να του δώσετε ζωή του θέματος αυτού. Και ε, σας ευχαριστώ πολύ όλους και για εσάς ε, κύριε κυρίες και κύριοι για τις παρεμβάσεις σας. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Να κάνουμε μισή ώρα διακοπή θα έλεγα. Θα επανέλθουμε στις 5.30 όπου έχουμε τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ, τα ξαναλέμε αργότερα. Stars en is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 Είναι να Yeah.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 Λοιπόν, παρακαλώ καθίστε. Λοιπόν, να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ε, μόνο ένα θέμα έχουμε. Οι προδιαγραφές για την υποδοχή ατόμων που αιτούνται διεθνούς προστασίας. Recast. Ο εισηγητής ε, ήταν ο κύριος Φέιν. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Λοιπόν, να σας αφήσω λίγο καιρό για τους τελευταίους που ορμάνε προς τις θέσεις τους. Για να μπορέσουν να βάλουν και στο μηχάνημα τις κάρτες τους. Οπότε, να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 93 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 94 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Συγγνώμη, 18, 18 υπέρ κατά. Να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Και εδώ ε, νομίζω ότι είναι αμφίβολο το αποτέλεσμα, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Δύο ψήφοι παραπάνω. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά Λοιπόν, ας ελέγξουμε και εδώ. Πέρασε. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Τέσσερις ψήφοι, πλειοψηφία. 21 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 97 όχι καταπίπτει 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική G υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε και εδώ γιατί είναι και συμβαστική πέρας εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. 100 υπέρ. Κατά. Λοιπόν, και εδώ να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται δύο ψήφοι περισσότερες υπέρ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί αρκετές τροπολογίες ε, δεν είναι αποδεκτές. Ah, sorry. Le 102. Η 102, 102 υπέρ, στη δεύτερη σελίδα, On vote le 102. Ψηφίζουμε την 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26. 26. υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Οπότε εδώ προχωράμε πιο κάτω. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική όμικρον ήταν αυτή. Τροπολογής 33, 130, 131 και 132 μαζί είναι ίδιες υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να τα πολιτεύσουμε, ήταν πολύ σαφέ. Μαζί 137, 138, 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατό 142. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36, ε, συγγνώμη, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 146. Να ελέγξουμε την 36. Δεύτερο τμήμα της 36. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας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 να ελέγξουμε την 152 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ίσα ίσα. 38, 153 και 154 μαζί. Υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, ψήφισα λάθος. Ήμουν υπέρ, όχι κατά. Αυτό θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Ε, πολύ αργά, λέει ο Πρόεδρος. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Δεν μπορούμε δυστυχώς να το αλλάξουμε. «38, 153 και 154 μαζί υπέρ» κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε 38, 153 και 154 μαζί. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνονται. Κύριε Πρόεδρε, να ζητήσουμε να λένε τσεκ μόνο τα μέλη, όχι βοηθή. Δεν είναι δική τους ευθύνη να λένε τσεκ για το ΕΛΚ. Το λέω. Ναι, πράγματι, μόνο οι βουλευτές μπορούν να ζητήσουν έλεγχο ηλεκτρονικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. 39, 155 και 156 μαζί υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά από, εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42, 168 και 169 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική έλα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά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 αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε τη 46 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με, κατά δύο ψήφους. 1 ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ...186 υπέρ... ...κατά... απόχέ. ...εγκρίνεται... ...187 υπέρ... ...κατά... απόχέ. ...εγκρίνεται... ...συμβιβαστική α... Συγγνώμη. 190 πρώτα απ' όλα. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική α αιτιολογική σκέψη ε, και υπάρχει προφορική τροπολογία, κύριε Μπενφέη. Ναι, έχουμε μία πρόταση της Άλντε. Ναι. ναι. Θέλουμε μια προταση της αλντε θελουμε μια προφορικη ε, τροπολογία μετά από το ensuring να ακυρώσουμε το all applicants are equal treated και να δικαταστήσουμε με standardized reception conditions for all applicants. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Αν όχι, να ψηφίσουμε την συμβιβαστική α. Ποιο είναι υπέρ, ποιο είναι κατά, αποχές, ε, γκρίνεται. Β. Συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Amendement 3 Τροπολογία 3 και 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ συγγνώμη καταπίπτει 55 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογίες 7, 60 και 59 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 61 υπέρ. Να ελέγξουμε τις 7, 60 και 59 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ α, καταπίπτει συγγνώμη 62 καταπίπτει 63 επίσης καταπίπτει πάμε στην 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 και 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Συμβιβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78, 79 υπέρ. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Καταπίπτουν 78 και 79. Πάμε στο 80. Υπέρ. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16. Ε. ξαναρχίζουμε, 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κα, κατά αποχές να ελέγξουμε να ελέγξουμε την 85 έρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται κατά μία ψήφο Υπήρχε λόγος να ελέγξουμε λοιπόν. 17-18 όχι. Πάμε στην 88 υπέρ. Κα... Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92 92 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ονομαστική με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας έγκρινεται συγχαρητήρια στον κύριο Σιγητή. Voilà, nous avons terminé, nous nous de... Ολοκληρώσαμε, θα βρεθούμε αύριο το πρωί στις 9.